Α Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση. Α, ε, ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, κύριε Νιούτον Ντάνα, από ό,τι βλέπω, είσαι ο μόνος βουλευτής που είναι παρόν σήμερα στην αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να πω ότι Κοιτάξτε, αυτό είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στου δικού μα θεσμού. είναι 9 και 20 και λαμβάνοντα υπόψη ότι χθε είχαμε την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και πάρα πολύ, από την Επιτροπή αυτή ή και τη δική μας είναι και μέλη της ΛΥΜΠΕ, άρα καταλαβαίνετε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι η συνέχεια των εργασιών ε, της χθεσινής και της προχθεσινής ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά και ομολογώ ότι νιώθω και πολύ δυσάρεστα απέναντι στους ε, καλεσμένους μας ε, για το ότι όσοι εδώ θα έπρεπε να είναι σήμερα στην ώρα τους έδειξαν έλλειψη, έδειξαν ανευθυνότητα. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι ε, να είχαν φτάσει κανονικά. Οι ε, οικοδεσπότες φτάνουν πριν από τους ε, καλεσμένους. Ehm, λοιπόν, ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και θέλω να κάνω μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση που αφορά στην παρέμβαση σήμερα το πρωί του Ιρλανδού Υπουργού, ο οποίος ε, μόλις πριν από λίγο μας είπε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει. Κατόπιν τούτου ε, δεν μπορεί σήμερα το πρωί να είναι εδώ στις εργασίες της ε, συνεδρίασής μας. Γι' αυτό λοιπόν αναθεωρήσαμε λιγάκι το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Και κατόπιν τούτου αναθεωρήσαμε και τον χρόνο αγόρευσης για το δεύτερο για τη δεύτερη ομάδα ε, θεμάτων, εκεί που γίνεται λόγος για την ε, συνεργασία κατά της νομοποίησης ε, εσόδων από κλιματικέ ενέργειε. Υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε γύρω στο 12, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και λίγο πιο πέρα. Ναι. Και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και αργότερα στη συνεδρίαση των συντονιστών. Στις 5.30 σήμερα το απόγευμα, στις 5.30 θα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ε, πρώτο θεματολόγιο που αφορά στην ε, ανακύκλωση ε, στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και στην ε, δέσμευση λογαριασμών. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω τη στρατηγική σημασία που έχει αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη μια εμπειρία για αυτό το θέμα και η εμπειρία αυτή μας δείχνει ότι κάτι που το επισήμαν άλλο και πάρα πολλοί δικαστές και πολλοί ερευνητές, ότι η κράτηση είναι αναμφίβολα η φυλάκιση, είναι ε, ένα από τα πιο αποτρεπτικά στοιχεία για τους ε, εγκληματίες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι και η δική τους υπερούσια Η περιουσία τους ε, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για κοινωνικούς σκοπούς. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι εγκληματίες έχουν παράνομα προσποριστεί περιουσιακά στοιχεία με βία, με καταχρήσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να τους αφαιρείται και να επιστρέφει στο, στους πολίτες σε, για κοινωνικούς σκοπούς. Θα έχουμε λοιπόν το Πέντρο Γκομές Περέρα, ο οποίος είναι ειδικό ε, από το Ινστιτούτο της ε, Βασιλείας, ε, Ινστιτούτο Διακυβέρνησης και η ομιλία του ε, φέρει τον τίτλο «Η ανάγκη για μια νέα ενωσιακή νομοθεσία που θα επιτρέπει στις, ε, στα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικέ ενέργειες να χρησιμοποιούνται για την κοινωνία των πολιτών και κυρίως για κοινωνικούς στόχους». Επίσης θα έχουμε και τον εκπρόσωπο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για τον εντοπισμό και την κατάσχεση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων αυτών, δηλαδή που έχουν προκύψει από εγκληματικές ενέργειες. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Περέιρα, ο οποίος ε, θα μιλήσει για ένα τέταρτο και επόμενος ομιλητής επίσης για ένα τέταρτο και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Περέιρα. Σας ευχαριστώ κύριε Λεφάνο, πρόεδρε της Ειδικής Επιτροπής. Scusi, signor Pereira, 30 eh, minuti. Ok, grazie. 30 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να καλώσω καλημερίσω όλους όσους είναι παρόντες ε, σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι παρόν ε, σήμερα εδώ για να παρουσιάσω τα αποτελέσματα και τις συστάσεις της μελέτης που έχει ο τίτλο ότι η ανάγκη για νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να επιτρέπει τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δημευτεί από τις εγκληματικές οργανώσεις να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνία των πολιτών και συγκεκριμένα για κοινωνικούς σκοπούς που υλοποιήθηκε από το Ιστιτούτο της για τη Διακυβέρνηση για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εισαγωγικά θα ήθελα να αναφέρω ότι ε, το Ίδρυμα είναι ένα εξάρτητο think tank χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς και επικεντρώνεται σε τομείς πρόληψης και καταπολέμησης διαφθοράς και νομοποίησης παράνομων εσόδων. Ιδρύθηκε το 2003 από τον καθηγητή Μάρκ Πιέθ ε, και το Ίδρυμα αναγνωρίζεται από τη γνώση και την εμπειρία του στους τομείς ε, της τεχνικής βοήθειας στη διαδικασία ανάκτησης περιοχής στοιχείων στην ε, δικαστική ε, συνεργασία και στην οικονομική έρευνα σε σχέση με τον εντοπισμό των προϊόντων και οργάνων του εγκλήματος. Υλοποιεί έρευνες και παρέχει συμβουλές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος και τα σχετικά συναφή εγκλήματα. Και η χρηματοδότησή μας προέρχεται από τις κυβερνήσεις του Λιχτεστάιν, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας. προκειμένου να εισαχθεί το θέμα της επαναχρήσης, της κοινωνικής επαναχρήσης των κατασκευμένων αγαθών, θα έπρεπε να ε, αναφέρω τη διαδικασία ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων. Γενικά η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο προέρευνας αναφέρεται στον εντοπισμό των πηγών πληροφοριών για να καθορίσουμε αν ε, έχει προκύψει ένα έγκλημα που πρέπει να ερευνηθεί. Δεύτερο στάδιο αναφέρεται στη συλλογή περιουσιακών στοιχείων και των απαραίτητων στοιχείων για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα αρμόδια άτομα, του αυτούργους, στο στάδιο αυτό που γίνεται η οικονομική έρευνα για να καθορίσουμε ποια είναι τα όργανα και τα προϊόντα του εγκλήματος προκειμένου να ζητηθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή η δέσμευση αυτών προκειμένου ε, να να μπορέσουμε να διακόψουμε την οικονομική ροή ε, προς τους δράστες. Τρίτο στάδιο έχουμε την ποινική διαδικασία κατά των αυτοργών και να ζητούμε την καταδίκη του. Στο στάδιο αυτό έχουμε την δίμευση των προϊόντων και οργάνων του εγκλήματος και τέλος, τέταρτο στάδιο, έχουμε την ανάκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων όπου ε, με δικαστική ε, εντολή γίνεται η ανάκτηση των χρημάτων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει ένα εύρωστο σύστημα αποφάσεων πλαίσεων και συνθήκων ε, σε σχέση με αυτά τα τέσσερα στάδια που αποτελούν τη διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ε, όμως, πρέπει να αναθεωρηθούν ε, οι πολιτικές της για να είναι πιο κατάλληλες ε, για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Βλέπουμε όμως, ωστόσο, ότι στην διαδικασία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν βλέπουμε άλλα δύο ουσιαστικά στοιχεία για την εν λόγω διαδικασία. Είναι η διαχείριση των κατασκευμένων στοιχείων, των δημευμένων αγαθών και η τελική, ο τελικός τους προορισμός. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς αφού έχουν κατασχεθεί πρέπει να εγγυηθούμε πώς χρησιμοποιείται καλύτερα αυτό το αγαθό. Το αντικείμενο της ε, μελέτης, ε, δηλαδή κοινωνική χρήση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται στον τελικό προορισμό αυτών των ε, στοιχείων, αυτών των αγαθών. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή ρυθμίση που να επιτρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιείται μία μεθοδολογία που επικεντρώνεται σε μία μελέτη προκαταρκτική που προέκυψε από ένα ερωτηματολόγιο που εστάλθηκε και στην κοινωνία των πολιτών αλλά και στα κράτη-μέλη. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την υλοποίηση αυτή της μελέτης ήταν να καθοριστούν οι όροι κοινωνική επαναχρησιμοποίηση και κοινωνικού σκοπή. Αυτοί οι όροι σήμερα δεν έχουν οριστεί και Όπως ε, θα φανεί από αυτή την παρουσίαση, αυτοί οι ορισμοί ερμηνεύονται γενικά αόριστα στα διάφορα κράτη-μέλη. Για τη μελέτη αυτή αναλύθηκαν ε, τα ακόλουθα σημεία κλειδιά. Καταρχήν, τα νομικά πλαίσια των ε, κρατών μελών με τα νομικά του συστήματα και τις πρακτικές, ε, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ανάκτηση περισσοϊκών στοιχείων. Αυτή η ανάλυση προσπάθησε να αναζητήσει την φυστάμενη νομοθεσία σε επίπεδο τοπικό και κοινοτικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επαναχρησιμοποίηση, κοινωνική επαναχρησιμοποίηση των περισσοϊκών στοιχείων. Το θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης αναλύθηκε για να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τον τελικό προορισμό αυτών ε, των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων στα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο των ε, θεσμικών πλαισίων ε, των κρατών μελών προσπαθήσαμε να καθορίσουμε τον κοινωνικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία αυτά και τέλος προσπαθήσαμε να καθορίσουμε ποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η παρουσίαση θα επικεντρωθεί λοιπόν στο θέμα που προτείνεται, την κοινωνική επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δημευθεί επικεντρωνόμενοι σε κάποιε εμπειρίε των κρατών μελών, ε, ακόμη και αν δεν υπάρχει ακόμη σε αυτά τα κράτη-μέλη ένα ορισμό τη ε, κοινωνική επαναχρησιμοποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορε αποφάσει πλαίσιο του Συμβουλίου σε σχέση με την ανάκτηση περιουσιακού στοιχείου, κυρίω σε ό,τι αφορά τη δέσμευση ε, αγαθών που είναι προϊόντα εγκλήματος ε, και ε, μπορεί να έχουν επιλεχθεί, να έχουν αναμειχθεί, να έχουν μεταπηθεί καθώς ε, και η δίμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν διάφορες μελέτες ε, και στρατηγικές που ασχολούνται με το θέμα της ε, δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, όμως το οργανωμένο έγκλημα πέρα από το ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές έχει και ένα κοινωνικό κόστος είναι σημαντικό ε, να αναφέρουμε την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί αναφέρεται ότι η επαναχρησιμοποίηση των ε, αγαθών που έχουν δεσμευτεί για κοινωνικούς σκοπούς προωθεί ε, μια στρατηγική καταπολέμηση του οργανωμένου έγκληματος ε, καθώς αυτά τα αγαθά θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα πόρος που έχει αφαιρεθεί από μια εγκληματική οργάνωση για να δοθούν επίσης ως ένας επικοδομητικός ε, παράγοντας που χρησιμοποιείται και στην πρόληψη του οργανωμένου κλίματος και στην πρόθεση την οικονομική και κοινωνική, της, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Όμως όσο δεν υπάρχει ρύθμιση για την ε, τολικό προορισμό των περιουσιακών στοιχείων αυτών ή για την επικοινωνική τους χρήση, Αφενός δεν υπάρχει αυτή η ρυθμισή, από την άλλη όμως υπάρχει ε, ουσιαστικά κάποιες πρωτοβουλίες για τον καλύτερο συντονισμό της νομοθεσίας ε, των κρατών μελών, έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους στο θέμα της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων. Επειδή δεν ε, υπάρχει ε, τέτοια ρύθμιση σε Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τα θέματα αυτά στην εσωτερική του νομοθεσία πως ο συντονισμός μεταξύ μελών, κυρίως στα πλαίσια του οργανωμένου εγκλήματος, θα εξαρτηθεί από ε, μια, έναν κατά περίπτωση ορισμό από τη χρήση της εσωτερικής νομοθεσίας των εμπλεκόμενων κρατών. Σε αυτή τη μελέτη έχουν ε, αναλυθεί έξι κράτη-μέλη δεν έχω χρόνο ούτε τους απαραίτητους πόρους για να κάνω μια πλήρη ανάλυση όλων των κρατών μελών. Αυτά τα έξι κράτη-μέλη που έχουν επιλεχθεί ήταν η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη η οι χώρες αυτές ε, επιλέχθηκαν ε, σύμφωνα με τα ακόλουθα προκαθορισμένα κριτήρια. Υπάρξη νομοθεσία για τη διαχείριση των δεσμευμένων αγαθών, η ύπαρξη σχετικών θεσμών για την ε, διαδικασία ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπω, ε, παραδείγματο χάρη η υπηρεσία ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπω προβλέπεται στην απόφαση 2007-845 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομικό σύστημα των κρατών μελών και οι ανάλογε πολιτικέ οργανώσει, ο ρόλος αυτών των κρατών μελών ε, στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η ποιότητα και αξιοπιστία των ε, στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, η προσβασιμότητα στις πληροφορίες και επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών και μια διαφορεμένη παρουσίαση εκπροσώπηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα επικεντρωθώ στη Βουλγαρία και στην Ιταλία που είναι τα δύο κράτη-μέλη τα οποία έχουν την ε, πιο προηγμένη νομοθεσία σε σχέση με την κοινωνική χρήση ε, των ε, περιουσιακών αυτών στοιχείων για κοινωνική χρήση. Η Βουλγαρία έχει ένα υψηλό ποσοστό οργανωμένου εγκλήματος. Για το λόγο αυτό οι βουλγαρικές αρχές έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το σύστημα δέσμευσης και δίμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως και της διαχείρισης αυτών αναζητώντας έτσι αποτελεσματικού τρόπους να εξουδετερωθούν τον οργανωμένο έγκλημα σε αυτή τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδη ο νόμος της απώλειας ε, προς όφελος του κράτους ε, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί ε, από εγκληματικές δραστηριότητες ουσιαστικά καταρχήν η διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ε, αναλαμβάνεται ε, από την αρμόδια υπηρεσία και καμία αρχή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να πουλήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Εδώ μιλώ για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλό κόστος ε, για το κράτος τη στιγμή της δέσμευσης και δίμευσης των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει κόστος για το κράτος γιατί πρέπει να διατηρήσει, να συντηρήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Και σε γενικές γραμμές ε, είναι μια αρμόδια υπηρεσία που αναλαμβάνει τη διαχείριση αυτών. Όταν ε, λοιπόν έχει γίνει δίμευση, περνούν στην κατοχή του κράτους, ε, το οποίο τα αναθέτει ουσιαστικά ε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα δεν υπάρχει ορισμός ε, κοινωνική χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτό ε, το νομοσχέδιο ε, προβλέπει τη δημιουργία ενός ε, ε, Συμβουλίου για τη διαχείριση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών που θα έχει την ευθύνη να προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών το να δορηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή να προτείνει την πώλησή τους. Και σύμφωνα πάλι με το νομοσχέδιο αυτό, πρόσωποι της Εθνικής Ένωσης ε, των Δημάρχων, των Δήμων, στη Βουλγαρία, οργανώσεις ε, μη κερδοσκοπικές και επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να κληθούν στις συνεδριάσεις αυτού του Συμβουλίου. Η μελέτη ε, βασίστηκε στο νομοσχέδιο όπως ήταν στην εκδοχή του Μαΐου του 2011. Το 2012 ήδη έγινε μια τροποποίηση αλλά είναι μόνο στα βουλγαρικά διαθέσιμα και εμείς ε, δεν ε, μπορέσαμε να συναντηθούμε με για να την αναλύσουμε. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει κάποιες συνεντεύξεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με τις βουλγαρικές αρχές και μας είπαν ε, ότι αυτό το τελευταίο στοιχείο θα είχε αφαιρεθεί και θα επέτρεπε σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ε, να συμμετάσχουν σε αυτό το Συμβούλιο. Και τέλος, σύμφωνα με το εν νομοσχέδιο, τα προϊόντα που προκύπτουν από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν μευθεί πηγαίνουν σε ένα ταμείο που το διαχειρίζεται ένα διοικητικό συμβούλιο και χρησιμοποιούνται οι πόροι για κοινωνικούς σκοπούς. Όπως παραδείγματο χάρη χρηματοδοτούνται ε, ταμεία κοινωνικής αρρωγής και προωθούνται μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Ε, στο βουλγαρικό παράδειγμα, όταν λέμε για κοινωνικούς σκοπούς, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε δραστηριότητες που αναπτύσσονται από το κράτος υπέρ της κοινωνίας, όπως ε, πολλές φορές... Ε, όπως φάνηκε και στο νομοσχέδιο, όταν ε, γίνεται λόγος ε, για ανθρωπιστικούς ε, λόγους, ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρήση και κοινωνικούς σκοπούς. Τώρα, η Γαλλική Δημοκρατία αναθεώρησε τον ποινικό κώδικα τον Ιούλιο του 2010 ε, για να διευκολύνει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Δημιουργήθηκε υπό την υποπτία του Υπουργείου Δικαιοσύνη και Υπουργείου Οικονομικών η Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάκτηση ε, των ε, δημευμένων και δεσμευμένων αγαθών. Αυτή η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και ως γενικός ε, κανόνας ο ε, ιδιοκτήτης ή ο πραγματικός δικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτών και μόνο σε ειδικέ περιπτώσεις ε, τα περιουσιακά στοιχεία θα τεθούν υπό ε, την εποπτεία αυτής της υπηρεσίας. Ο στόχος εδώ είναι ουσιαστικά να υπάρχει μεγιστοποίηση τη αξία των περιουσιακών στοιχείων υποδήμευση. Οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα δεν περιλαμβάνουν κάποιες διατάξεις για την τελικό προορισμό των ε, αγαθών αυτών των περιουσιακών αυτών στοιχείων ή ε, δεν καθορίζονται κάποιες αρχές που εμπλέκονται. Έτσι λοιπόν, οι διαδικασίες αυτές στη Γαλλία υπάρχουν ε, στη περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται με περιπτώσεις ε, διακίνησης ναρκωτικών. Στις δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των ε, προϊόντων του εγκλήματος ε, για χρήση για την κοινωνία των πολιτών. Αν και μπορούμε να καταλάβουμε ότι ε, το ταμείο αυτό που υπάρχει και γίνεται κατάσχεση του περισσοτικού στοιχείων των προϊόντων διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιούνται οι πόροι για να βοηθηθούν οι τοξικομανείς. Στην ε, γαλλική περίπτωση γίνονται κάποιες προσπάθειες την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε μία περίπτωση του σε, ε, υπόθεσης bien mal acquis, δηλαδή περισσότερο στοιχείο που έχει αποκτηθεί διά της ε, πλαγίας οδού. Εκεί είχαμε μία απόφαση του κυρωτικού δικαστηρίου για να ουσιαστικά διερευνηθεί μια καταγγελία που είχε γίνει από ενώσεις ε, καταπολέμησης της διαφθοράς. Στην ε, περίπτωση αυτή, αν μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία για κοινωνικούς σκοπούς, θα ενίσχυε ένα σύστημα πιο αντιπροσωπευτικό και διαφανής και θα διευκόλυνε μια συμμετοχή πιο δραστική της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τώρα, να συνεχίσουμε με την Ιταλική Δημοκρατία. Η Ιταλική Δημοκρατία είναι σήμερα η μόνη χώρα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ειδική νομοθεσία που αναφέρεται στην διάθεση των ε, κατασκευμένων περιουσιακών στοιχείων και κοινωνικού σκοπού. Η Ιταλική νομοθεσία καθορίζει ότι ορισμένα είδη περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα λόγου χάρη, διαβιβάζονται προς, μια κοινό, προς την κοινότητα όπου δημεύτηκαν για να χρησιμοποιηθούν για την τοπική κοινωνία, για, κάποιες για κάποιους ή ενώσεις. Το 2010 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε Εθνική Υπηρεσία για τη Διαχείριση και το τελικό προορισμό ε, των ε, περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασκευθεί από το οργανωμένο έγκλημα προκειμένου ε, να η υπάρξει διαχείριση αλλά και μελλοντική διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μετά τη δίμευσή τους. Η υπηρεσία ε, διαθέτει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε τοπικές κοινότητες ή ε, σε επαρχές για να επαναχρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν υπό την ιδιοκτησία δημοσίων αρχών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα σχέδια ή είναι αντικείμενα διαχείριση από τρίτου, όπω το χάρη από την κοινωνία των πολιτών, οργανώσει κοινωνία πολιτών, χωρί κερδοσκοπικού σκοπού. Εδώ παρουσιάστηκε ο βασικός ε, μηχανισμός ε, στο ιταλικό μοντέλο, σας το εξήγησα μόλις, και πρέπει να τονίσουμε ότι ισχύει μόνο για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, παίρνουμε τους χαρτών, μιλάμε για σπίτια ή για άλλα κίνητα, για άλλες ιδιοκτησίες. Και όταν μιλάμε για κινητά αγαθά, παραδείγματος χάρη για τραπεζικούς λογαριασμούς ή ε, για κάποια περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες ή αλλού, αυτά, αυτή η αξία δεν ε, πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται για κοινωνικούς σκοπούς αυτά τα ποσά η υπηρεσία διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων ε, από νομικά πρόσωπα Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 η υπηρεσία είχε αποδώσει 87,1% των απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες αρχές, σε κοινότητες και σε ε, επαρχίες, συνομαρχίες επίσης, γίνεται και μία παρακολούθηση της διαχείρισης ε, στη συνέχεια αυτών των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να μην υπάρξει δίσδυση στη διαχείρισή τους από το οργανωμένο έγκλημα και παρακολουθείτε για το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Η υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα, την εξουσία να ανακαλέσει την μεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή να διορίσει έναν ειδικό επίτροπο. Αν διαπιστώσει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα, να περάσουμε στο γερμανικό μοντέλο. Η Γερμανία, όπως ε, είδαμε και στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Γαλλίας, ουσιαστικά ε, καλύπτει την, ε, κάποιες υποχρεώσεις του αστικού κώδικα. Πρόκειται για ένα ομοσπονδιακό σύστημα εδώ και επομένω ε, δεν υπάρχει μία και μόνη υπηρεσία για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Ε, αρμόδιο είναι το κάθε λέντε. Το κάθε Στην περίπτωση της Βάδης Βιτεμβέργης, Αυτό το κρατήδιο έχει συγκεκριμένες υπηρεσίες για τη δέσμευση και, την και τη δέσμευση και τη δίμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε αστυνομικούς αλλά και δικαστές που είναι αρμόδιοι. Στο σημερινό σύστημα τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία πηγαίνουν στον προϋπολογισμό του κρατηδίου όπου είχαμε την ε, πρώτη δίκη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε δραστηριότητα που προβλέπεται στο προϋπολογισμό. Μπορεί να υπάρχει βέβαια και μια κοινωνική πτυχή εδώ, όμως δεν είναι η χρήση που έχει δηλωθεί για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην ε, Βρέμη προβλέπεται ένα τμήμα ε, των περιουσιακών στοιχείων αυτών να ε, πάνε στο γερουσιαστή, στη γερουσία για τη δικαιοσύνη και για το Σύνταγμα και επίσης ένα άλλο τμήμα, 24.000 ευρώ, για τον τομέα της εργασίας νεολαία προστασία των γυναικών κτλ. Για να κατεπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων και για να βοηθηθούν οι τοξικομανείς. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει μία ε, κοινωνική χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όμως το κράτος είναι αρμόδιο για την εποπτεία αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Περνάμε τώρα στο ισπανικό μοντέλο και αυτό το μοντέλο μοιάζει με το γαλλικό, το βουλγάρικο και το γερμανικό. Δεν υπάρχει ένα καθεστώ διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και η διαχείριση καθορίζεται από κάθε δικαστή αναπερίπτωση. Η αξία του ισπανικού μοντέλου είναι ότι υπάρχει ένας ε, θεσμικός μηχανισμός που ε, μας επιτρέπει οποιοδήποτε πολίτης, είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, να ε, μπορέσει να κάνει μια καταγγελία προκειμένου να υπάρξει έρευνα από τις Ισπανικές Αρχές. Στην περίπτωση αυτή για την ε, χρήση των περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικό στόχο θα μπορούσε η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει με πιο δραστικό τρόπο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και τέλος, έχουμε το βρετανικό μοντέλο εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός που λέγεται Community Cashback, όπου τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία επανεπενδύονται υπέρ της κοινότητας περίπου 95.000 λίρες ε, χρησιμοποιούνται ε, υπέρ των κοινοτήτων. Η κοινωνία γενικά μπορεί να παρουσιάσει κάποια σχέδια, κάποια project για χρηματοδότηση μέσω συνεδριάσεων με την τοπική αστυνομία. Γίνονται κάποιες συνεδριάσεις σε τοπικό επίπεδο με τις τοπικές αρχές. Ο στόχος θα ήταν ε, να αποκτήσουν μεγαλύτερη φωνή οι τοπικές κοινότητες για το πώς θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν και να επανεπενδυθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στις τοπικές κοινωνίες. Την περασμένη Παρασκευή έχουμε μαθεύτηκε κάτι που αναφέρεται στη Σκοτία και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη χρήση αυτών των αγαθών που είναι οι εξοδικαστικές συμφωνίες σε αυτό το μοντέλο, στην περίπτωση της Σκοτίας, το Abbott Group συμφώνησε, ο Όμιλος Abbott, ε, δημιούργησε μία συμφωνία με τον ε, εισαγγελέα της Σκοτίας ότι πρέπει να πληρώσει 5 εκατομμύρια λίρες, μία αξία, ένα ποσό που ε, ουσιαστικά φαίνεται ότι η επιχείρηση απέκτησε μέσω διαφθοράς για ε, να χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό για κοινωνικούς σκοπούς υπέρ των νέων. Για μια ακόμη φορά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει συνιστόσα του κοινωνικού σκοπού. παρόλα αυτά το κράτος είναι αρμόδιο για τη διαχείριση αυτών των αγαθών. Αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Από ό,τι βλέπω έχω μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή μου. Η σημερινή ρύθμιση δεν μας ενημερώνει το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία κατόπιν την ε, αποκτησή τους από το κράτος. Επίσης, η κοινωνική επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι μία κοινή πρακτική στα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αναγκαιότητα να συζητηθούν τα πλεονεκτήματα ε, για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για κοινωνικούς σκοπούς. Έτσι όπως ε, μας εξήγησε και η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωμοδότηση που αφορά την εσωτερική ασφάλεια, οι τοπικές κοινότητες είναι αυτές που πληρώνουν το πιο υψηλό τίμημα του οργανωμένου εγκλήματος ε, και η κοινωνική επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων υποδήμευση θα μπορούσε να αποζημιώσει τις ε, κοινότητες αυτές που έχουν πληγεί η επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικού σκοπού επιτρέπει στι τοπικέ αρχέ που έχουν πληγεί από το οργανωμένο ή σοβαρό έγκλημα να είναι σε καλύτερη θέση για να καταπολεμήσουν το έγκλημα αυτό. Το να επιτρέψουμε την συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων όπω και στην ίδια την ανάκτηση στη διαδικασία ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Επίση, μα επιτρέπει να αυξήσουμε την δράση εκ των προτέρων ε, τη ε, κοινωνία των πολιτών στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του σοβαρού και του οργανωμένου κλίματο. Και αν μου επιτρέπετε να μου δώσετε τρία ακόμη λεπτά, θα ολοκληρώσω. Να αναφέρω ως παράδειγμα της ε, αποτελεσματική καταπολέμησης από την πλευρά τη κοινωνία των πολιτών και το πώς θα μπορούσε να ευνοηθεί. Εγώ αναφέρω όχι μόνο την περίπτωση της Γαλλίας που ακούσατε πριν, αλλά και μια περίπτωση στην Ισπανία, όπου η κοινωνία των πολιτών προέβη σε μια δράση για να διερευνηθεί η υπόθεση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ε, ε, σε σχέση με την υπόθεση των Μπακ στην ε, σημερινή Γουινέα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι για να ενισχυθεί το ίδιο το δικοστικό σύστημα των κρατών ε, προκειμένου να είναι πιο δημοκρατικά και επίσης ε, προκειμένου και να εκπαιδευτούν οι πολίτες ε, στο πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επειδή δεν έχω χρόνο, Νομίζω ότι σε όλα αυτά που ανέφερα και στον ορισμό και στις δυνατότητες που υπάρχουν, να σας πω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με τις εξοδικαστικές συμφωνίες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ ενό κράτου και ενό ιδιώτη, πώ θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για κοινωνικού σκοπού και ιδίω όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα διασυνοριακό. Τη στιγμή δηλαδή που καθορίζεται ποια είναι η κοινότητα θύμα, ποιο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή το κράτο που έχει στην κατοχή του ε, αυτά τα περισσοϊκά στοιχεία ή το κράτος που έκανε την έρευνα και έχει κατασχέσει αυτά τα περισσοϊκά στοιχεία. Αυτό το θέμα θα έπρεπε να μελετηθεί στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης, του τρόπου επαναχρησιμοποίησης αυτών των περισσοϊκών στοιχείων. Οι συστάσεις τώρα. Έχουμε τέσσερις ε, συστάσεις. Η πρώτη είναι να δημιουργηθούν διαφανείς διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση των δημιουργημένων περιουσιακών στοιχείων. Η οδηγία θα μας έλεγε υπό ποιες προϋποθέσεις τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για κοινωνικούς σκοπούς ε, τα κατασχημένα περιουσιακά στοιχεία ή θα μπορούσε ένα συγκεκριμένο ποσό να χρησιμοποιείται για κάθε κράτος μέλος ε, για κοινωνικούς σκοπούς ή ένα τμήμα αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ε, κατόπιν αποζημίωση των θυμάτων. Μια δεύτερη συστασία και δεν δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τα με τα σχεμένα περιουσιακά στοιχεία, αυτή η βάση δεδομένων θα επέτρεπε στα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να καθορίσουν τον τρόπο χρησιμοποίηση ε, των περιουσιακών στοιχείων αυτών, καθώ ε, εκεί θα είχαμε στατιστικά στοιχεία από τι αρμόδιε υπηρεσίε ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ε, που υπάρχει σε κάθε κράτο μέλο. Αυτή η σύσταση όμως θα ε, προσέθετε κάτι στις λειτουργίες αυτών των αρμόδιων υπηρεσιών. Τρίτη σύσταση θα ήταν η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ανάκτηση περιοσιακών στοιχείων. Θα δημιουργόταν ένα συγκεκριμένο ταμείο στο οποίο ένα μέρος της αξίας, της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων θα κατατεθόταν σε αυτό το ταμείο και κατόπιν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για ευρωπαϊκά project με κοινωνική συνιστόσα. Δηλαδή είτε εντό είτε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ είναι διασυνοριακό το οργανωμένο έγκλημα και μπορεί να υπερβεί τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και τέλο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρε σύστημα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ε, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που θα ήταν υπεύθυνη για να, δημιουργη... για να διασφαλίσει ότι σε όλε τι περιπτώσει, τι υποθέσει που έχουμε διασυνοριακό χαρακτήρα, θα υπάρχει παρακολούθηση από την υπηρεσία αυτή. Θα συνεργαζόταν με τι αντίστοιχε υπηρεσίε υπηρεσίες των κρατών μελών και θα διασφάλιζε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Το πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας, ενός ευρωπαϊκού γραφείου θα ήταν ότι θα είχαμε μια εναρμονημένη ερμηνεία ε, του όρου κοινωνική σκοπή. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Καλή θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, στον Ιάν Ντάβιτσον, ο οποίος θα μας μιλήσει για την Βρετανική εμπειρία, κυρίως ε, όσον αφορά ε, τον εντοπισμό και τη δέσμευση ε, προϊόντων εγκληματικών ενεργειών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλημέρα. Δεν είναι πολύ χρόνος το τέταρτο αυτό. ασχολούμαι και με την Αγγλία και με την Ουαλία και με τη Σκοτία. Και ολόκληρο δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ασχολούμαι όπως σας είπα και η Πρόεδρος με το θέμα μεταξύ άλλων του ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος και της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε εννέα ομάδες κατάσχεσης και δίμευσης και καθήκον τους είναι να διερευνούν όλα αυτά τα θέματα, κατασχέσεις, πλήσιμο κλπ. Στην Αγγλία και την Ουαλία βασιζόμαστε κυρίως, αλλά και στη Σκωτία. Όπως ξέρετε όμως στη Σκωτία υπάρχει διαφορετικό νομικό σύστημα, δικαστικό σύστημα. και ως προς τις δημεύσεις και κατασχέσεις. Σήμερα θα κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ αγγλικού και σκοτικού συστήματος. Θα προσπαθήσω να σας αναφέρω τα θετικότερα στοιχεία και από τα δύο. Δεν είναι εδώ θεωρητικές οι παρατηρήσεις αυτές, αλλά βασίζονται στην εμπειρία πολλών ετών. Ελπίζω να μπορέσω να σας εξηγήσω και τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία για να μάθετε από την εμπειρία μας. Πρώτον, να σας κάνω μία γενική επισκόπηση, παρουσίαση του, της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασίλειου. Πρώτον, η δίμευση, η κατάσχεση. Έπειτα, έχουμε το δικαίωμα να κατάσχουμε περιουσιακά στοιχεία παράλληλα με την ε, εγκληματολογική, με την ποινική δίωξη. Και αυτά τα χρησιμοποιούμε και μέσω της αστυνομίας και μέσω των γενικότερων δυνάμεων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Τα δικαστήρια μπορούν επίσης να αποφασίσουν δίμευση. Αν ένα άτομο πολύ μικρά, μικρές ποσότητες ναρκωτικών στον δρόμο πάλι μπορεί να οριστεί από δικαστήριο όμως η δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια ε, ο, ο βαθμός της κατάσχεσης ε, είναι σχετικός με, την, με το αδίκημα και με το κατά πόσον είναι γνωστός, εσημασμένος, κακοποιός ή όχι. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατακρατεί 50% όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων και το 12% του χρηματοδοτεί τις περιφερειακές ομάδες δίωξης του εγκλήματος. Και τα υπόλοιπα δίνονται αλλού. όταν κατάσχονται χρήματα πάλι κρατιέται το 50% από το Υπουργείο. ...18,7% χρηματοδοτεί στη Σκοτία το, τις διοκτικές αρχές, 18,7% στα δικαστήρια. Αυτά όλα έγιναν χωρίς καμία σωστή ανάλυση του πραγματικού κόστους. Αν θέλει κανείς να βρει κάποιον τρόπο αντικειμενικότερου καθορισμού αυτών των ποσοστών, ας το κάνει. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την προώθηση της, της δίωξης του εγκλήματος. Τα θετικά του αγγλικού συστήματος είναι ότι επιβραβεύει κατά κάποιον τρόπο την δίμευση, την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που να χρηματοδοτούν τη δίωξη. Έχουν υπάρξει πολλά θετικά παραδείγματα, όχι όμως όλα. Οι δημοσιονομικοί ελεγκτές βέβαια δεν ασχολούνται ειδικά με θέματα των κερδών από το έγκλημα αλλά ασχολούνται και με όλες τις ποινικέ διώξεις, εγκλήματα, δολοφονίες κλπ. Δεν είναι εύκολο να δούμε ποσοτικά πόσο ωφελεί αυτό τις διοκτικές αρχές. Ο προϋπολογισμός της δίωξης του εγκλήματος προωθείται πάντως και το Υπουργείο Εσωτερικών παραδέχεται ότι δεν είναι και τόσο διαφανή όλα αυτά. Από τα αρνητικά θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη στόχευση προς εκείνους που απειλούν περισσότερο την κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί οργανωμένοι εγκληματίες κρύβουν τα περιουσιακά του στοιχεία και δεν προκύπτουν πολλά από την κατάσχεση λόγω του πλησίματος βρωμίκου χρήματος. Και υπάρχει ο πειρασμός της ε, δίμευσης και κατάσχεσης που χρησιμοποιείται απλώς και μόνο για να μην αλλάξει τίποτε. Αυτό δεν είναι πολύ θετικό. το Υπουργείο Εσωτερικών ε, προσπαθεί να καθορίσει πόσα χρήματα χρειάζεται. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κύριος στόχος είναι να αφαιρεθεί, να σταματήσει η δραστηριότητα όσων είναι επικίνδυνη για την κοινωνία. Πιστεύω ότι αν η ιδεοντολογική προσέγγιση γενικευόταν, τότε θα καταλήγαμε σε περισσότερα κέρδη από τις κατασχέσεις. γιατί υπάρχει ο κίνδυνος οι κατασχέσεις να καταλήξουν σε μεγαλύτερη προώθηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να συνεννοηθούμε λοιπόν με τους ακαδημαϊκούς. Η αναγνώριση των κινδύνων που εγκυμονεί η προσέγγιση του κυνηγήματο των περιουσιακών στοιχείων είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί όλα τα σώματα δίωξης του εγκλήματος δεν μπορούν να βασίζονται για τη λειτουργία τους στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών γιατί έτσι μπορεί να καταλήξουν να είναι μια κερδοσκοπική οργάνωση και δραστηριότητα αντί της αγνής δίωξης. Στο βιβλίο του The Laundryman ο Τζέφρι Ρόμπινσον από το 1994 αναγνώρισε ότι κύριο στόχος δεν πρέπει να είναι οι δημεύσεις και τα κέρδη από αυτές αλλά η ακριβώς η δίωξη του εγκλήματος. Αν τέτοιοι στόχοι γενικεύονταν, δηλαδή οι δημεύσεις κατασχέσεις και τα κέρδη από αυτές, τότε δεν θα υπήρχε σε λίγο αστυνομία, θα ήταν απλώς ένα κερδοσκοπικό σύστημα. Γι' αυτό το εγγλικό σύστημα μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί η ιδεοντολογική ή η ηθική προσέγγιση να παραγραφεί τελείως. Το σύστημα δεδομένων, συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει ομάδες και άτομα για να γίνεται πιο εύκολα η έρευνα. Τουλάχιστον 30% των εγκληματιών έχει αποδειχθεί ότι τα κέρδη τους τα δαπανούν άμεσα για να μην αφήνουν ίχνη. Άρα δεν μπορούμε να ερευνήσουμε το οργανωμένο έγκλημα με βάση την έρευνα των περιουσιακών του στοιχείων, γιατί υπάρχει το πλήσιμο. Βέβαια η νομοθεσία για την καταπολέμησή του υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν λοιπόν ωφέλη, υπάρχουν και κίνδυνοι. Εάν η χρήση των κατεσχημένων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι διαφανής. Το σκοτσέζικο μοντέλο τώρα ήταν και είναι διαφορετικό. Πριν το 2010 όλα τα κατασκευμένα στοιχεία επέστρεφαν στην κοινότητα με βάση το πρόγραμμα Cashback for Communities. Υπάρχει όμως πίεση και στη Σκοτία να χρησιμοποιηθούν οι κατασχέσεις με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Αγγλία. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατασχέσεις για τη χρηματοδότηση διάφορων δραστηριοτήτων όπως του κοριτσίστικου ποδοσφαίρου και άλλα τέτοια. Είναι φανερό ότι τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις. Υπάρχει και πρόγραμμα χρηματοδότησης νεανικού μπάσκετ. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι μπορούν πιο άμεσα να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη αυτά για κοινοτικέ δραστηριότητες και αποδεικνύουν ότι είναι αποτελεσματική επικοινωνιακά τουλάχιστον η δίωξη του εγκλήματος. Και έτσι δεν υπάρχει και ο κίνδυνος να πούμε ότι η αστυνομία θα κυνηγάει πάντοτε την κερδοφορία αντί την απλή δίωξη του εγκλήματος. στο Εδιμβούργο εδρεύει η βασική μονάδα χρήσης αυτών των κατεσχημένων περιουσιακών στοιχείων. Φαίνεται όμως ότι οι επενδύσεις σε τοπικά προγράμματα δεν ήταν ούτε εκεί ακριβώς αυτές που θα μπορούσαν να είναι ή θα έπρεπε να είναι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός δημοσιονομικός ελεγκτής για κάθε τέτοια δραστηριότητα. Στη Σκωτία όμως δεν υπάρχουν τέτοιοι τοπικοί επόπτες ή ελεγκτές. Γι' αυτό έγινε μία έρευνα σε τρεις τοπικά αστυνομικά τμήματα στις χειρότερες εγκληματικές περιφέρειες και φάνηκε ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων δεν στόχευε πάντα όσο δυνατόν καλύτερα τη χρήση. Με συγχωρείτε αλλά τα λέτε πολύ γρήγορα. Οι μεταφράστριες δεν προλαβαίνουν. Λοιπόν. Αν αλλάξει αυτό το... Είτε μπορεί να γίνει καλύτερη στόχευση και αύξηση των κατασχέσεων. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι φανερό τι πρέπει ακριβώς να γίνει στη Σκοτία καθώς θα συνδυάζονται οι διοκτικές αρχές μεταξύ τους. Πάντως καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και πιο συνδυασμένα όλα αυτά. Ποιο είναι τα μαθήματα λοιπόν. Το αγγλικό σύστημα έχει ορισμένα θετικά στοιχεία αλλά δυστυχώς ε, έχει και αρνητικές επιπτώσεις ενώ το σκοτσέζικο χρησιμοποιεί άμεσα τα χρήματα για κοινοτικούς σκοπούς αλλά τελικά μπορεί να μην του στοχεύει πολύ καλά. Υπάρχει ο πειρασμός η χρησιμοποίηση των δεδημευμένων περιουσιακών στοιχείων να μην καταλήξει σε πρόοδο της δίωξης. Στην Αγγλία έχουν γίνει προσπάθειες οι κατασχέσεις να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο ή δείκτης της αποτελεσματικότητας της δίωξης, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. γιατί η καλή χρήση των ε, κατεσχημένων δεν είναι ο κύριος στόχος μας που είναι η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Εμείς θέλουμε να καταστραφούν οι δραστηριότητες αυτές. Πολλές φορές η κατάσχεση μερικών εκατοντάδων λιρών από κάποιο διαρρήκτη δεν έχει το ίδιο βάρος με την κατάσχεση χιλιάδων λιρών από ένα οργανωμένο δίκτυο και επομένως μπορεί το ποσό που κατάσχεται να μην είναι σοβαρός δείκτης της σοβαρότητας του εγκλήματος. Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι έχουν φέρει ορισμένα αποτελέσματα, αλλά το αγγλικό πρόγραμμα κινήτρων ίσως δεν έχει χρησιμοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Φαίνεται ότι και τα δύο προγράμματα έχουν κάποια θετικά στοιχεία η βασική αρχή πρέπει να είναι ότι όλα τα κατεσχημένα στοιχεία πρέπει να επιστρέφουν στην κοινότητα τους. Μπορούν να εξισορροπηθούν τα δύο σχήματα, προγράμματα. Και η επαναχρησιμοποίηση των ποσών αυτών για την προώθηση των δραστηριοτήτων των διοκτικών αρχών δεν είναι κακό στοιχείο αλλά δεν πρέπει να περιορίζεται η δραστηριότητά τους στις κατασχέσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά και για εκπαιδευτικά προγράμματα και με την καταλληλότερη χρήση της τεχνικής που επιτρέπει ο νόμος, αλλά πρέπει όλες οι διοκτικές αρχές να επιδιώκουν και πρόσθετη χρηματοδότηση και χρήση πιο ειδικευμένων εποπτών και ελεγκτών. Με προτεραιότητες βέβαια. Τέτοια επενδυτικά προγράμματα μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει πρώτα να υπάρξει ανάλυση του κινδύνου που είναι η στόχευση κυρίως των χρημάτων και των κατασχέσεων δεοδός δεν θα έπρεπε να επιστρέφουν τέτοια χρήματα στην κυβέρνηση, αλλά μόνο στην κοινότητα ή στη χρηματοδότηση των ίδιων των διοκτικών αρχών. Μπορεί να γίνει καλή τους χρήση, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται πάντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε να εκφράσω και εγώ κάποιες απόψεις. Ε, και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος ε, Φερέιρα ο οποίος ε, είπε ότι είναι απαραίτητο να επαναχρησιμοποιούν ε, τα κατασκευθέντα αυτά αγαθά προς όφελος ε, της κοινωνίας. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές ακριβώς τις, αυτόν τον καιρό δουλεύει πάνω σε μια οδηγία για, τις, για την κατάσχεση. Δυστυχώς βέβαια η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει απολύτως τίποτα για την επαναχρησιμοποίηση. Εγώ, και άλλοι στην Επιτροπή ε, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή τη πολύ μεγάλη έλλειψη γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, δηλαδή είναι τεράστιο το κόστος για τα κράτη για τη διαχείριση των αγαθών ε, και τη συντηρησή τους. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ε, ήρθαν ε, επαφής με μένα διάφορες δικαστικές υπηρεσίες οι οποίες διαμαρτύρονται και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρουν και αυτοί που διαχειρίζονται τα αγαθά. Ε, όλοι λοιπόν αυτοί επισήμαναν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν τα αγαθά αυτά με την πραγματική τους αξία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κατά νου. Διότι αν είναι αλήθεια ότι πρέπει να ε, δούμε λιγάκι και να υιοθετήσουμε τις ε, πιο προχωρημένες νομοθεσίες άλλων κρατών μελών. Από την άλλη βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε να ξαναπέσουμε στα ίδια λάθη, δηλαδή να επανέλθουμε σε καταστάσεις οι οποίες θα απαγορεύσουν μια θετική αναθεώρηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιακολίνο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το θέμα της ε, δίμευσης, ε, είχαμε τους ε, δύο μιλητές οι οποίοι τοποθετήθηκαν για το θέμα αυτό και εσείς επίσης το ίδιο και είναι σαφές ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να εγκριθεί στο Κοινοβούλιο η πρόταση οδηγίας. Βεβαίως καλύπτοντας ε, το κενό ε, το οποίο αναφέρατε. Οι δύο μιλητές αναφέρθηκαν στο ιταλικό μοντέλο αυτό της ε, Βουλγαρίας και υπάρχουν και άλλα όπως αυτό της Ισπανίας που αξίζει τον κόπο να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Ινστιτούτο Δέσμευσης ε, το ε, υπερεθνικό είναι πολύ σημαντικό, ε, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάσχεση και την διαχείριση αυτών των αγαθών. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να καθορίσουν ένα κείμενο το οποίο θα προβλέπει ακριβώς την επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικούς ε, σκοπούς και θα προβλέπει επίσης ε, ότι από τη στιγμή που έχει κατασχεθεί ή δημευτεί ε, η περιουσία, τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στο κράτος. Άρα δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει ακόμα με πιο αποτελεσματικό τρόπο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτά τα εγκληματικά προϊόντα. Υπάρχει δηλαδή η δίμευση και μετά πρέπει να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτόν τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιακολίνο και τώρα εκ μέρους της άλλου του κύριου Νιούτον Ντάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να διαβεβαιώσω και τους δύο ομιλητές ότι ακόμα και αν πολλά μέλη είναι σε άλλες επιτροπές, ό,τι και αν μας πείτε, εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ ε, χρήσιμο και θα καταγραφεί στα πρακτικά μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, τα άδεια έδρανα δεν είναι και τόσο σημαντικό. Βεβαίως ζητώ συγγνώμη που είναι άδεια. Μία ερώτηση προς τον κύριο Περέιρα καταρχήν. Μήπως υπάρχει ένας διεθνής μηχανισμός που να μπορεί να ε, ορίζει όταν υπάρχει κατάσχεση σε διεθνές επίπεδο, ποιος παίρνει τα κατασχεθέντα ή μήπως τσακώνονται οι κυβερνήσεις η μία να λέγω θα πάρω 50% και εσύ άλλο το 50%. Υπάρχει ένας ε, μηχανισμός για τέτοιου είδου ε, περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλό ότι το διεθνές έγκλημα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Και μία άλλη ερώτηση θα ήθελα να μας πείτε το εξής. Τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε το χειρότερο παράδειγμα όπου ε, τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά και να πρέπει να το έχουμε κατά νου, γιατί θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Και κάτι άλλο, ε, εσείς έχετε μελετήσει και την Αμερική, γιατί έχετε ασχοληθεί κυρίως με την Ευρώπη. Έχετε μήπως και κάποια εμπειρία από την Αμερική. Και προς τον κύριο Ντέιβιτσον τώρα επειδή μιλάμε οι την ίδια μετρική γλώσσα, νομίζω ότι οι λέξεις που ε, επιλέξατε ήταν πολύ προσεγμένες και θα ήθελα να έχω κι άλλη μια κατηδίαν συνάντηση με εσά ε, για να μάθω περισσότερα. Είπατε ότι δαπανάνε τα χρήματα, ε, τα, το προϊόν εγκλήματος, πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πιει υπερβολική σαμπάνια, υπάρχει κάποιο όριο. Και αν αγοράσουν σπίτια, αυτά θα κατασχεθούν. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η ταχεία διασπάθηση του χρήματος. Και κάτι άλλο. Προς τον κύριο Chris Mathers, Ε, μπήκα στο Google και δεν τον βρήκα. Δεν ξέρω μήπως δεν έγραψα καλά το όνομά του. Ποιο είναι το όνομα του συγγραφέα και πώς λέγεται το βιβλίο που πρέπει να διαβάσουμε. Ευχαριστούμε, Μπιλ. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψει να δώσω εγώ έτσι μια πρώτη απάντηση. Δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί με τα χρήματα ε, που ε, προσπορίζονται. Πριν από λίγο καιρό, εδώ στις Βρυξέλλες, η Ντράγκετα αγόρασε σε τέσσερις ώρες 28 εκατομμύρια ευρώ. Αγόρασε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο μέσα σε ελάχιστες ώρες. Βλέπεις λοιπόν πώς μπορούν να κινηθούν. Ε, ο κύριος Ματία, παρακαλώ, για να απαντήσει. Με συγχωρείτε, κυρία Ματία. Ματία. Ευχαριστώ. Μπορώ να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είδαμε στην γαλλική τηλεόραση της προάλλες ότι η μαφία δανείζει σε, με τεράστια επιτόκια σε φτωχούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη και αντικαθιστά τις τράπεζες. Έτσι λοιπόν ε, αποκτά μεγάλο έλεγχο του πληθυσμού σε πολλές χώρες. Και εγώ ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τον πρώτο, από τον πρώτο μιλητή. Κύριε Περέιρα, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την παρέμβασή σας, ε, γιατί είχα λιμένες υποχρεώσεις, άλλη συνεδρίαση, αλλά η συνεργάτες μου πήρε σημειώσει. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω ε, τα όσα προτείνατε. Να ρωτήσω τον κύριο Ντέιβινσον. Ελπίζω να μπορείτε να μου απαντήσετε. Γνωρίζετε περιπτώσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη δίμευση περιουσιακών στοιχείων Δηλαδή όχι σε περίπτωση που να έχουμε ποινική καταδίκη, αλλά καταδίκη βάση του αστικού δικαίου. Γνωρίζετε κάποια περίπτωση σχετικά με το αν ε, ο ύποπτος ε, αθωώθηκε ε, και τι έγινε στη συνέχεια με τη δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. Γιατί έχουμε κάποιες πολιτικές διαφωνίες με την Επιτροπή είτε στο Συμβούλιο είτε στο Κοινοβούλιο για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και κατόπιν ε, για να συμφωνήσω με την κυρία λοιπόν είμαστε πολύ που η πρόταση της Κομισιόν δεν περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία δηλαδή για τον προορισμό αυτών των ε, περιουσιακών στοιχείων. Τελικά έχουμε μία μισή πρόταση της Κομισιόν, γιατί ωραία, κατάσχουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μετά τι τα κάνουμε. Ελπίζω να μπορέσουν να προτείνουν κάτι παραπάνω, αλλά δεν ξέρω αν η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να, δεχτούν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Κυρία Βάλερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να επανέλθω στην πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα ε, το Κοινοβούλιο να συμπληρώσει την ε, πρόταση αυτή, δηλαδή με την έννοια ότι μπορούν να υπάρχουν αποκεντρωμένα κοινωνικά προγράμματα τα οποία ενδείκνυνται έτσι ώστε τα κατασχεθέντα είτε είναι κινητέ, είτε είναι ακίνητες εξίε, να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικού σκοπού. Νομίζω λοιπόν ότι την πρόταση Κομισιόν μπορούμε να την εμπλουτίσουμε και αυτό το έχουμε κάνει πολύ συχνά. Εγώ έχω μία ερώτηση που αφορά ε, σε αυτά που ρώτησε ο συνάδελφος ε, Νταν. Ε, ρώτησε για την εμπειρία από τι ΗΠΑ και θέλω να ρωτήσω μήπω και στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει μια υπηρεσία που να επιλαμβάνεται του θέματο αυτού. Γιατί μπορώ να φανταστώ ότι ε, κάποιοι εγκληματίες ε, δεν ε, βρίσκονται στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική αλλά σε κάποιες, κάποια κακόφημα νησιά και τις δουλειές τους τις κάνουν μέσα από το διαδίκτυο. Μήπως υπάρχουν λοιπόν οι δομές εκείνες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο να τους εντοπίσουμε. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξή. Γνωρίζω ότι στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η διαδικασία μέχρι να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης ε, με το να μπορεί κανείς να διαχειριστεί ελεύθερα ε, τα κατασκευτέντα. Και στην Ιταλία είδαμε ότι επικρατεί μία νεφελώδης κατάσταση. Οι υπηρεσίες δεν δίνονται να διαχειριστούν τα χρήματα κατατοδοκούν γιατί ενδέχεται να πρέπει να επιστρέψουν κάποια ποσά αν τελικά ε, το, η δικαστική διαδικασία καταλήξει αρνητικά για το κράτος. Έχετε λοιπόν εσείς πληροφορίες ε, για την ταχύτητα ή για φραγμούς, δηλαδή αν μια διαδικασία, μια υπόθεση ξεπεράσει το χρόνο, νομίζω αυτό δημιουργεί πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση. Δύο λεπτά, ο κύριος Μπορσελίνο. Η κυρία Μπορσελίνο. Κοιτάξτε, από ό,τι άκουσα, ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση, ε, περιεκτική, ασχολήθηκε με όλες τις ε, αποχρώσεις του θέματος και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί πραγματικά ε, συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες του κυρίου Αλφάνο αλλά και άλλων ε, συναντέλφων που μίλησαν πριν από εμένα. Θα ήθελα λοιπόν δυστυχώς λέω δυστυχώς, να αναφερθώ στην Ιταλική νομοθεσία. Η Ιταλία είναι πρωτοπόρα σε αυτό το θέμα γιατί εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με το θέμα. Όπως ε, ξέρετε έχουν ε, ε, υπάρξει στην Ιταλία πολλά τέτοια σοβαρά σημαντικά θέματα. Η Ιταλία λοιπόν θεωρώ ότι έχει ποσοτικά πολύ περισσότερα τέτοιου είδου κατασκευαίνοντα προϊόντα από ότι άλλε χώρε. Η εγκληματικότητα σε εμά ε, διαρκεί εδώ και πολύ καιρό και άρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσχεση ποσοτικά είναι μεγάλη. Επίσης, ε, οι περιουσίες που έχουν κατασχεθεί μπορεί να μην είναι όλες μεγάλες, μπορεί να είναι κατατμημένες, πιο μικρές. Είναι λοιπόν δύσκολο, ειδικά αυτές οι μικρές, ε, να ε, χρησιμοποιηθούν. Και θέλω λοιπόν γι' αυτό το λόγο να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Να πω το εξής. Στην Ιταλία έχουν αρχίσει να μιλούν για την κατάσχεση ενός μαφιόζου, ο οποίος όμως ε, δολοφονείται. Μιλάμε, αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 και την αναθεώρηση περί ε, διαχείρισης πάνω στοιχείων την είχαμε δεκαετία του 90. Είχαμε λοιπόν μια μακρά περίοδο όπου η Ιταλία έκανε την εμπειρία ότι όπου ε, η περιουσία δεν μπορούσε να την διαχειριστεί το κράτος. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ε, τα οποία εντωμεταξύ βέβαια έχασαν την αξία τους, ε, ήταν αντικείμενο βανδαλισμού. Κατόπιν τούτου, εγώ θεωρώ για άλλη μια φορά ότι αυτή η Ιταλική εμπειρία μπορεί να χρησιμεύσει έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι αποφάσεις που Δυστυχώς, ε, από ό,τι φαίνεται, δεν προβλέπεται τέτοια ε, ρύθμιση στην πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άκουσα λοιπόν να γίνεται λόγος για κάτι πολύ σημαντικό για την Τράπεζα Ενδομένων, αλλά και ένα είδος ταμείου. Ένα ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται κυρίως τα αγαθά εκείνα που είναι δύσκολο να είναι αντικείμενο διαχείρισης όσον αφορά την πώληση. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα γιατί μπορούν να περάσουν στην περιουσία των ε, μαφιόζων αλλά τουλάχιστον να πολλούνται κάποια αγαθά έτσι ώστε να μπορεί να συντηρείται και το ταμείο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να υπογραμμίσουμε την ε, χρησιμοποίηση αυτών των αγαθών, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το ηθικό μήνυμα που εκπέμπεται. Η μαφία δεν θα πρέπει να μπορεί να πει ότι ε, τα χρήματα τα οποία είχε ήταν ε, στα χέρια της μαφίας παραγωγικά και μάλιστα στα χέρια του κράτους γίνονται και βάρος για τους πολίτες. Αυτό δεν πρέπει να μπορεί να το ισχυριστεί η μαφία. Αυτό εξάλλου είναι και το μήνυμα της μάχης κατά της ε, μαφίας. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω ε, το λόγο στους ε, φιλοξενούμενους μας για να απαντήσουν. Κύριε Περέρα, ξεκινώ με εσάς. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομος για τους διεθνείς μηχανισμούς. Με ρωτήσατε αν υπάρχουν για τη δίμευση και για την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων σε διμερές επίπεδο υπάρχει. Υπάρχει στη Σύμβαση των Ηνωμένων κατά της διαφθοράς η πρόθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε αυτή τη σύμβαση, είναι μέρος αυτής της σύμβασης, αλλά υπάρχουν και διμερείς συμφωνίες έτσι ώστε κάθε κράτος να επιλύει ε, τον τρόπο που θα διαχειριστεί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, του πώς θα το κάνει. Υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο. Τώρα, τα αφιαλτικά σενάρια υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ να σας πω, ως παράδειγμα, μια υπόθεση όπου είχαμε κατάσχεση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού, δύο δισεκατομμύρια δολάρια, και όλα αυτά ήταν σε επενδυτικά ε, ταμεία, σε επενδυτικά κεφάλαια. Η ερώτηση είναι πώς διαχειρίζεται το κράτος ένα επενδυτικό κεφάλαιο. Δεν έχει ικανότητα, δεν έχει αρμοδιότητα το κράτος, δεν έχει ειδικού εμπειρογνώμονες για να κάνει επενδύσεις σε μετοχές ε, και σε άλλα προϊόντα. Οι εγκληματίες δαπανούν πολύ γρήγορα χρήματα και μάλιστα και με μοναδικά πράγματα. Εγώ γνωρίζω περιπτώσεις με το χάρη ένα άτομο είχε ένα ζωολογικό κήπο. Θα ε, ήθελα να σας ε, ρωτήσω, ένας εισαγγελέας, ένας δικαστής, ξέρει ε, πόσα κιλά κρέας είναι μια καμιλοπάρδελη που πρέπει να, ή πόσα κιλά κρέας πρέπει να φάει ένα λιοντάρι, ξέρει πόσο κοστίζει η συντήρηση του ζώου αυτού. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και γι' αυτό εδώ το πράγμα της Ιταλίας ε, ξέρω ότι και η Κολομβία έχει παρόμοια προβλήματα με τη διακίνηση ναρκωτικών. Μιλάμε για υψηλό κόστος, δηλαδή να διατηρηθεί η παραγωγικότητα όπως γίνεται με μια επιχείρηση. Πώς γίνεται αυτό. Υπάρχουν ε, διάφορα μοντέλα, ήταν και μία από τις ερωτήσεις αυτές για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Μπορούμε να διατηρήσουμε όπως το βρετανικό ή το γαλλικό μοντέλο, να υπάρχει συντήρηση ε, του περιουσιακού στοιχείου, να, το, να διατηρείται αυτό ως εγγύηση ενώ μία άλλη λύση θα είναι να ε, μπουν, να ρευστοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να μπουν σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο που μου δώσατε, όμως να δώσω και μια τελευταία απάντηση. Αν υπάρχει κάποιος άλλος οργανισμός, ε, νομίζω ότι ρώτησε η κυρία Βάιλερ από τη Γερμανία, αν ε, τα Ηνωμένα Έθνη αν στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει ε, ένας οργανισμός που να συνεργάζεται ε, με περιφερειακές οργανώσεις ε, σε άλλους σε πιο τοπικό επίπεδο. Ναι, υπάρχει στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κ. Ντέβιτσον για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτο ερώτημα. Πώς δαπανούν τα λεφτά τους οι εγκληματίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούμε ως εγκλημα, οργανωμένο έγκλημα ακόμη και απλούς λοποδίτας και λοποδίτριες. Μπορεί λοιπόν να δαπανίσουν τα χρήματά τους οποτεδήποτε και οπωσδήποτε και μετά να συνεχίσουν να εγκληματούν. Όσο για το βιβλίο του Χρήστου Μάιδερς, το έχω αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει γι' αυτό. Αυτά που είπε η κυρία Μάθιου για δημεύσεις ή κατασχέσεις μετά από αστική αγωγή. Αυτά αφορούν κυρίως ανθρώπους που έχουν πεθάνει, ή έχουν φύγει από τη χώρα και όπου δηλαδή υπάρχει επαρκής απόδειξη, εφόσον υπάρχει επαρκής απόδειξη εγκληματικής δραστηριότητας ή προέλευσης των χρημάτων. Είναι δεν έχω όμως καμία εμπειρία από συγκεκριμένες περιπτώσεις αν πέτυχε ή απέτυχε η κατάσχεση, δεν μπορώ να σας πω. Όσο για την εμπειρία των ΗΠΑ, έχω επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως με το FBI και είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Εκεί υπάρχει πολύ ομοσπονδιακό επίπεδο δίωξης παραπάνω από ό,τι σε μας εδώ στην Ένωση και εκεί έχουν κατασχέσει εκατομμύρια εκατομμύριων δολαρίων αεροπλάνα, ιδιωτικά κλπ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στο ομοσπονδιακό επίπεδο είναι πολύ δυνατή, αλλά στο τοπικό βέβαια μοιάζει με εμάς. Όσο για οργανωμένες μεθόδους κατασχέσεων δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο α, χρειάζονταν κατά μέσο όρο 22 μήνες για κατάσχεση μετά από καταδίκη. Φαντάζεστε αν προσθέσουμε 2-3 χρόνια για την ίδια την έρευνα και το χρόνο που θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί η απόφαση βλέπετε πού φτάνουμε οι πιο πολύπλοκες περιπτώσεις και που αποφέρουν περισσότερα σε εισαγωγικά κέρδη είναι γνωστές αλλά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες που έχουν παραμείνει άγνωστες. Η Ιταλική εμπειρία είναι ενδιαφέρουσα και συμφωνώ με τη δεοντολογία της. Όσο για την τράπεζα δεδομένων για τις κατασχέσεις, ή ανακτήσεις, Έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια τέτοια εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πρέπει να ενημερωθεί. να ε, τη εφαρμοστεί ένα σύστημα καλύτερης διαχείρισης, δηλαδή γιατί έχουν γίνει πολλά λάθη. Ελπίζω να απήντηστα. Ευχαριστούμε κυρία Ντέβιτσα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη συνεισφορά σας για ένα ζήτημα που όπως ε, είδατε και από τη συζήτηση είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολεί τα μάλα. Θα σας ζητούσα να αφήσετε στη γραμματεία της Επιτροπής μας ε, την παρέμβασή σας, ε, αλλά και οποιαδήποτε περαιτέρω ιδέα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στις εργασίες μας. Τώρα, θα ήθελα να καλέσω εδώ στο βήμα τον κύριο Μαν Σερβίζη. Παρακαλώ. Είχα μια ερώτηση για τον κύριο Γκόμες Περέιρα. Δεν ε, ξέρω πότε πρέπει να θέσω αυτή την ερώτηση, αλλά Θα μπορούσα να τη θέσω τώρα. Okay. So, well, I'll Θα μιλήσω πορτογαλικά. και αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Εμεί εργαστήκαμε στα πλαίσια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την έκθεση Μακοβέη που αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ε, μέσω της Δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από κλιματικές δραστηριότητες. Συγγνώμη που έφτασα αργά, όμως με ενημέρωσαν για την παρέμβασή σα και μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς. Όπως στην Ιταλία υπάρχουν εμπειρίες ανάκτησης ε, και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υπέρ των θυμάτων Ίσως ε, θα μπορούσατε να μας ε, δώσετε κάποιες ε, περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το ταμείο, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να συσταθεί και ποιοι οργανισμοί, ποιοι θεσμοί θα έπρεπε να συμμετέχουν εκεί, τι κοινοβουλευτικό έλεγχος θα μπορούσε να υπάρχει και ποια πρόσβαση θα μπορούσε να υπάρχει, και όχι μόνο από την πλευρά των θεσμών, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. Και ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η ιδέα δημιουργίας του Ταμείου θα ήταν βάση της ε, εμπειρίας ε, στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το community cashback, δηλαδή ένα ποσοστό αυτό, της αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων να πήγαιναν σε αυτό το ταμείο, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες των θυμάτων, αλλά και η, την ίδια, την η ίδια κοινωνία των πολιτών από τις κοινότητες αυτές θα μπορούσε να προτείνει κάποια project και θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, Ευρωπαίοι ελεγκτές ε, για το μηχανισμό αυτό. Αυτό το ταμείο πιθανότατα, συγγνώμη δεν θυμάμαι ε, το όνομα στα πορτογαλικά, αλλά είναι η γάμα δέλτα ιστορικών υποθέσεων. και θα μπορούσε να συμμετέχει εκεί και η Europol και άλλοι μηχανισμοί. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Περέιρα. Τώρα, κάλεσα προηγουμένω στο βήμα εδώ του Προεδρείου τους ομιλητές για το επόμενο κλάστερ. Ε, θα ακούσουμε στο δεύτερο κλάστερ που αφορά την ενίσχυση του πλαισίου για αποτελεσματική διασυνοριακή δίμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Θα ακούσουμε τον κύριο Μεσερβίση, ο οποίος είναι Γενικό Διευθυντής της ΓΑΜΑ Ιστορικών Υποθέσεων, που θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της δίμευσης των περιουσιακών στοιχείων. Κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μίλ Βαντερντό από την Παγκόσμια Τράπεζα που θα μα μιλήσει για τα εμπόδια στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τι διεθνεί εξελίξει στον λόγο τομέα. Θα δώσουμε 15 λεπτά σε κάθε ομιλητή και κατόπιν το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, κύριος Μανσερβίση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα, γιατί θεωρώ πάντοτε ότι αυτή η Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για την όθηση και την υποστήριξη ε, για πρωτοβουλίες που έρχονται που δεν έρχονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι λοιπόν πραγματική ικανοποίηση και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Να σας πω ότι χαίρομαι που βλέπω ότι υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν για την ε, δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. Είναι φεδαζωτική υποστήριξη αυτή και είναι κατανοητό. Ε, ασκείται για κάποια κριτική, αλλά νομίζω ότι είναι καλό το ότι όλοι θέλουμε να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν θέλω να με κρηγορήσω, να σας πω που βρισκόμαστε σε σχέση με το νομικό πλαίσιο, τα γεγονότα και κατόπιν να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για τις δραστηριότητες τις ε, ευρύτερες, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την νομοθεσία εδώ. Κάποια γεγονότα. Γνωρίζετε βέβαια τα πράγματα καλύτερα από ότι εγώ το οργανωμένο έγκλημα, επιδιώκει το κέρδος, έχουμε πάρα πολύ υψηλά αριθμητικά στοιχεία. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι η γνώση των όταν δεν είναι ερμονισμένη, δεν έχουμε λοιπόν στην πραγματικότητα μία ε, σαφή και κοινή εκτίμηση για το πόσο τεράστιο είναι το φαινόμενο αυτό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε κάποια νούμερα που μας δίνουν κάποια κράτη-μέλη. Στην Ιταλία συγκεκριμένα 150 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 και είμαι σίγουρος ότι είναι και υποεκτίμηση αυτή. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε επίσης για κάποια δισεκατομμύρια, αλλά ποσοτικά είναι τεράστιο το φαινόμενο. Αλλά να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ποσότητας αλλά και ποιότητας. Το οργανωμένο έγκλημα είναι διεθνές, είναι διασυνοριακό και όσο πιο ολοκληρωμένε είναι η οικονομία μας, δείτε την ενιαία αγορά. Αλλά δείτε και τι πρόκειται να κάνουμε προκειμένου να απαντήσουμε στην οικονομική κρίση, τη μελλοντική τραπεζική ένωση, την δημοσιονομική ένωση κτλ. Ε, όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, αν δεν ε, συνοδεύεται από συμμετρικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, όλα αυτά οι και σίγουρα στο μέλλον θα δουν δίσδυση του οργανωμένου κλίματος. Έχουμε ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό που θέλω να υπογραμμίσω και φυσικά θα πρέπει να δοθούν περισσότερες προσπάθειες εκεί για το ότι είναι διασυνοριακό αυτό το έγκλημα και εκμεταλλεύεται πλήρως ε, όλες τις δομές της παραοικονομίας. Η τρίτη πτυχή είναι ότι μπροστά σε αυτό το τεράστιο ποσοτικό φαινόμενο και το ποιοτικά σημαντικό, το αποσά και τα περιουσιακά στοιχεία υποδήμευση είναι σχετικά μικρά, ούτε εδώ έχουμε αρμονισμένα νούμερα, αλλά όσα έχουμε μας δείχνουν ότι στην πραγματικότητα αυτές οι δραστηριότητες ε, παραμένουν ένα ποσοστό του φαινομένου. Τώρα, αυτά είναι κάποια γεγονότα. Να σας πω τώρα που βρισκόμαστε στο νομικό πλαίσιο. Η δική μας αξιολόγηση, η δική μας εκτίμηση ήταν, γι' αυτό προτείνουμε συγκεκριμένη οδηγία, ότι δεν επαρκούν τα σημερινά μέσα. Η οδηγία πλαίσιο δεν εφαρμόζεται πλήρως καταρχήν. Δεύτερον, είναι πολύ αόριστη και δεν μας επιτρέπει να έχουμε αποτελεσματική δράση σε δικαστικό επίπεδο και σε επίπεδο διοκτικών αρχών, κυρίως ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των διασυνοριακών υποθέσεων. Επομένως, διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, είναι αρκετά χαλαρό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως προκύπτει αναγκαιότητα να κάνουμε περισσότερα. Ο Μάρτιο υιοθετήσαμε μια πρόταση οδηγίας που επίσης προσπαθεί να απαντήσει στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οδηγία αυτή προσπαθεί να προσδιορίσει ακριβώς ε, ποια είναι τα κενά, τα πιο σημαντικά στη σημερινή κατάσταση και πολύ συχνά το περιθώριο της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Καταρχήν, υπάρχουν σαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά τη διευρυμένη δίμευση. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να δούμε σε ποιο περιβάλλον ε, εργάζεται, το λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα και να το κατεπολεμήσουμε. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διευρυμένη εικόνα και να έχουμε και διευρυμένη δίμευση φυσικά πάντα με τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες. Ε, η πρότασή μας προσπαθεί να δημιουργήσει αυτήν την ισορροπία. Έτσι λοιπόν έχουμε πρώτον ε, αυτή την διευρυμένη δίμευση και δεύτερον έχουμε τη δίμευση τρίτου μέρους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να αποφύγουμε τα αγαθά, τα περιουσιακά στοιχεία απλώς να μεταβιβαστούν σε ένα άλλο άτομο που δεν ε, ε, είναι κατηγορούμενο σε μια συγκεκριμένη ύποπτα, σε μια συγκεκριμένη έρευνα, αλλά θα μπορούσε να συμμετέχει στον οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή να λειτουργεί ως άτομο στον οποίο διατίθεται τα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ε, δίμευση χωρίς να υπάρχει καταδίκη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή σε ορισμένες περιπτώσεις, περιορισμένες περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε την ποινική καταδίκη, να μπορούμε να προβούμε σε δίμευση σε κάποιες περιπτώσεις, σε λίγες περιπτώσεις, όταν έχουμε θάνατο ε, του ατόμου αυτού ή όταν έχει διαφύγει ή όταν είναι άρρωστο το άτομο αυτό. Τέταρτον, να διασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές, όπως οι εισαγγελείς προσωρινά, να μπορούν να δεσμεύσουν προσωπικά στοιχεία που θα εξαφανιστούν αν δεν αναλυφθεί δράση. Έτσι λοιπόν μιλάμε εδώ για προληπτικές αρμοδιότητες δέσμευσης αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δεν μπορέσουμε να αδράξουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα εξαφανιστούν και θα εξαφανιστούν όχι απλώς σε μια χώρα, θα εξαφανιστούν ε, στην ενιαία αγορά ε, τουλάχιστον στην δική μας ολοκληρωμένη οικονομία. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε κοινού κανόνες γιατί διαφορετικά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια απόφαση για δέσμευση ε, που να εκτελείται ε, από διαφορετικές δικαστικές αρχές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Κατόπιν, πέμπτον, ε, η αστυνομία και οι εισαγγελίε μπορούν να συνεχίσουν τις έρευνες ε, για τα προσωπικά στοιχεία του καταδικαστέτα όταν έχει δοθεί εντολή για την κατάσχεση ενό συγκεκριμένου ποσού, αλλά δεν έχουν κατασχεθεί επαρκή περιουσιακά στοιχεία. Θέλουμε λοιπόν να πάμε εκεί όπου το κέρδο μπορεί να έχει μετατραπεί σε κάτι που δεν σχετίζεται άμεσα με το έγκλημα, αλλά σίγουρα σχετίζεται με το άτομο που ε, είναι ο δράστης. Θέλουμε δηλαδή ουσιαστική δράση που σε οποιαδήποτε περίπτωση θα μπορεί να ερευνηθεί από τους δικαστές και την αστυνομία. Υπάρχουν κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και απαιτούν από τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν κατάλληλα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, γιατί ξέρετε, η τεχνική της μαφίας είναι ακριβώ να φέρει αξία από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να τα ξαναγοράσει στη συνέχεια ή απλώ να δείξει ότι μόλι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ε, τελικά ε, αφαιρούνται από αυτούς, χάνουν και αξία. Επίσης, ε, θέλουμε εδώ να μην είναι το οργανωμένο έγκλημα πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση των περισσοικών στοιχείων. Αυτό είναι ένα από τα θέματα το, το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να το καταπολεμήσουμε. Και τελευταίο σημείο Δεν θα σας πω πολλά, αλλά όλοι αυτοί οι τομείς είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το τεκμηρίο της αθωότητας. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που θα προστατεύουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά προτείνουμε λοιπόν συνολικά. Τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω εις βάθος ε, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στις διαπραγματεύσεις, οργανικές διαπραγματεύσεις της οδηγίας. Και γιατί τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε μία συζήτηση και με τα κράτη-μέλη. Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Απλώς επιτρέψτε μου να πω από τη σκοπιά της Κομισιόν ότι Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία να φοβόμαστε ότι αυτή η προσέγγιση, η οποία αυτή καθευτεί, δεν είναι επαναστατική, γιατί πρέπει να εργαστούμε βάσει του άρθρου 83. Επομένω, πρέπει να κάνουμε κάποιε υποχωρήσει. Αλλά υπάρχει ένα κίνδυνο αποδυνάμωση και θα έχουμε δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό όταν θα, θα φτάσει η συζήτηση διοργανική στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά να σας πω ότι Δυστυχώς ε, δεν είναι και πολύ συναρπαστική. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα βιαστούμε προς το να βρούμε ένα κοινό παρανομαστή και αν ε, σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχουν ε, ε, ισχυροί κανόνε σε κάποια εθνική νομοθεσία, τότε θα στραφούμε προ τα εκεί. Όμω, εμεί δεν θέλουμε κατά τη δική μα προσέγγιση. Είμαστε πεπισμένοι ότι είτε θα έχουμε μια υψηλότερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή, ή ε, το απλό, αν κάνουμε ένα απλό patchwork ε, των διάφορων εθνικών νομοθεσιών, τότε θα επιτρέψουμε στο εργανομένο έγκλημα να εκμεταλλευτεί αυτές τις διαφοροποιήσεις και οι ιδιοκτικές ε, αρχές δεν θα μπορούν να συνεργαστούν κατάλληλα προκειμένου να καταπολεμήσουν το φαινόμενο. Πρέπει λοιπόν όλοι να επαγρυπνούμε γιατί όλα αυτά γίνονται με ένα πολύ τρόπο αλλά θέλω να ευστήσω την προσοχή σας σε αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια λεπτή στιγμή, δηλαδή πάντα θα υπάρχει η τάση να εξεύρουμε συμβασμό, γιατί δεν μπορούμε να συζητούμε και για χρόνια, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ λεπτό και σημαντικό ζήτημα και αυτό σχετίζεται και με την κατάσταση που ζούμε την οικονομική κρίση, δηλαδή την αγκαιότητα να προστατεύσουμε την ε, νόμιμη οικονομία, δηλαδή το δικαίωμα των ε, ανθρώπων να λειτουργούν νόμιμα, να δραστηριοποιούνται νόμιμα επιχειρηματικά. Και ξέρετε, το οργανωμένο έγκλημα είναι μια βιομηχανία και καθώς ε, εναρμονίζουμε τους κανόνες να επιτρέψουμε ε, στο νόμιμο κομμάτι να ε, μπορεί να δραστηριοποιείται στην ενιαία αγορά, πρέπει να κάνουμε και το ίδιο, να έχουμε κανόνες και νόμους για να αποτρέψουμε την παραοικονομία στην ενιαία αγορά τις παράνομες δραστηριότητες. Τώρα, οι δύο συνεδευτικές δραστηριότητες που είναι πολύ σημαντικές και τις έχετε σήμερα το πρωί, το ένα είναι η υπηρεσία, τα γραφεία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και το άλλο είναι η χρήση ε, αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Για το πρώτο, νομίζω ότι είναι μια δουλειά που προοδεύει. Η νομοθεσία έχει προβλεφθεί το 2009, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο τώρα το οποίο συνδέεται και με τη Europol και εργάζεται καλύτερα, λειτουργεί καλύτερα, αλλά είναι ένα δίκτυο που πρέπει να γίνει ακόμη πιο ενεργό, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Αν μπορούμε να συνεισφέρουμε κατά κάποιο τρόπο και με κονδύλια, ξέρετε, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και δραστηριότητες από αυτή τη σκοπιά. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε λοιπόν και σε αυτού και επίσης να υπάρξει και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή έχουμε τα κεντρικά μητρώα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ε, πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να ανταλλαγεί βελτιστών πρακτικών. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά πρέπει να δούμε πώς πρακτικά θα λειτουργούμε καλύτερα, όχι μόνο να μένουμε σε επίπεδο νομοθεσίας. Τώρα το δεύτερο θέμα αφορά τη χρήση των ε, κατασκευμένων περιουσιακών στοιχείων. Παρά τη βούλησή μας, δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε αυτό με την πρόταση που υποβάλαμε. Υπάρχει πρόβλημα με τη νομική βάση. Η νομική βάση είναι το άρθρο 83. Δεν ήταν δυνατό να καλύψουμε και αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε να φεύγουμε έναν τρόπο, να σκεφτούμε πώς ε, θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Είναι πρόβλημα της νομικής βάσης και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό δεν υπάρχει νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη ισοδύναμη, επομένως η βάση εναρμόνισης ήταν επίσης ε, αδύναμη. Και τι προτιμήσαμε να κάνουμε, να δώσουμε ένα συμβασμένο ότι αυτή είναι μία πορεία προς την οποία πρέπει να κατευθυνθούμε μαζί. Και γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα για κάποιου λόγους, όπως είπα στην αρχή, επειδή το οργανωμένο έγκλημα αποσκοπεί στο κέρδος, όσο χτυπάμε το κέρδος ε, τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε και επειδή υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες, ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα κράτη λειτουργούν, είναι καλύτερα από το έγκλημα. Έτσι λοιπόν, όταν κατάσχουν, όταν δημεύουν, περιουσιακά στοιχεία τα ξαναδούν στην κοινωνία και καθώ η μαφία δείχνει την ισχύ της, τον ελέγχει την επικράτεια, στον να ε, τους ανθρώπους, τους πολίτες, ότι όσο περισσότερο συμμετέχουν, ε, τόσο καλύτερο για αυτούς, σε εκείνες τις δομές, τους δείχνουμε ότι όχι. Τα κράτη είναι αυτά που δίνουν πίσω τα περισσότερα στοιχεία και δημιουργούν νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες. Πρέπει να εργαστούμε ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και εμεί είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σα και να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά σε αυτό το θέμα δεν υπήρχε νομική βάση. Τώρα, αυτή την app τη Σκοπιά, καλώ ορίζω ότι πρέπει η πλατφόρμα μα να δημιουργήσει μια υποομάδα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει το πώ μπορούμε να έχουμε έναν πιο κοινό πολιτισμό για να συγκρίνουμε νούμερα και στοιχεία και να προκύψουν κάποιε ιδέε. και αν μπορούμε να το συμπληρώσουμε αυτό με κάποιες συγκεκριμένε δράσει που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα μελλοντικά ταμεία, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε από αυτού. Δηλαδή βλέπουμε με σαφήνεια ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και είχα και την ευκαιρία να επισκεφθώ κάποια ακίνητα στην Απουλία που έχουν κατασχεθεί και ξαναχρησιμοποιήθηκαν για κοινωνικούς σκοπούς και μπορώ να σας πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε όχι μόνο ότι χρησιμοποιήθηκαν και πάλι για παραγωγικούς σκοπούς αλλά δόθηκαν πάλι στους πολίτες ε, και τώρα η μαφία έχει εξαπολύσει να επιτύχει και προσπαθεί ακριβώς ε, να διαλύσει αυτή την επιτυχία δείχνοντας ότι δεν παράγουν πλέον αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, καταστρέφουν ε, την παραγωγή της οικονομικής δραστηριότητας και καταστρέφουν και αυτή την πεποίθηση προκειμένου να προκαλέσουν διαταραχές στην κοινωνία. Αυτά τα σχόλια είχα, αυτές τις παρατηρήσεις είχα να κάνω και αυτά τα στοιχεία σας να σας υπενθυμίσω. Όπω σα είπα, πρέπει να συνεχίσουμε την κίνημα μα πορεία και να είμαστε και έτοιμοι για κάποιε σκληρέ διαπραγματεύσει, έτσι ώστε τελικά να έχουμε κάποια αποτελέσματα που θα μπορούν τουλάχιστον να συγκριθούν με το μέγεθο του προβλήματο που θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Διευθύντα. Και τώρα ο δόκτωρ Βαντερντούς από την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα μας μιλήσει για τους φραγμούς και τα εμπόδια στις ανασχέσεις και ανακτήσεις. Ορίστε κύριε μου. Πρόεδρε, εξοχότατα μέλη, Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Είμαι από τη μονάδα κατασχέσεων και ανακτήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και της αρμόδιας μονάδας του ΟΗΕ. Το 2007 σε μια προσπάθεια να συγκεκριμενοποιηθούν αυτά που λέγονται στο κεφάλαιο 5 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, όπου, καθορίζονται, όπου καθορίζεται η βασική αρχή της ανάκτησης, λέγεται ότι περιουσιακά στοιχεία που έχουν παρανόμως ε, κτηθεί πρέπει να, από κάποια χώρα πρέπει να επιστρέφουν σε αυτήν. Και το ΣΤΑΡ με τρεις τρόπους το πράγμα αυτό. Βασίζεται σε τρία εργαλεία. Πρώτον, είναι σημαντικό όσοι ασχολούνται με τις ανακτήσεις, δηλαδή οι διοκτικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές, οι αντιδιαφθορικές αρχές να έχουν την απαραίτητη γνώση, να ξέρουν πώς γίνεται ο δημοσιονομικός έλεγχος και πώς μπορεί να γίνει η ανάκτηση που ζητάει κάποια τρίτη χώρα. Να υπάρχει λοιπόν η γνώση και μία βάση δεδομένων, τεχνογνωσία. Αυτό είναι το πρώτο θεμέλιο. Έχουμε συγγράψει οδηγούς που αφορούν και τους πολιτικούς και τους ασχολούμενους με τη δίωξη πώς μπορεί καλύτερα να χρησιμοποιήσει κανείς τον αστικό κώδικα, τον ποινικό κώδικα και πώς γίνονται οι δημοσιονομικοί έλεγχοι, τι πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς από μια τράπεζα, τέτοιου είδους πρακτικά θέματα γράφουμε. Δεύτερο θεμέλιο, να διασφαλίσουμε ότι τα διεθνή πρότυπα που υπάρχουν η ειδική task force για τα δημοσιονομικά παραδείγματο χάρη εφαρμόζονται και ενδυναμώνονται και εφαρμόζονται από δικηγόρους, τράπεζες και, και από όποιον ασχολείται με ανακτήσεις για να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια των νομικών και δικαστικών δομών. Όταν υπάρχει μία προφανής περίπτωση διαφθοράς διαπλέκονται διάφοροι οργανισμοί εκεί μέσα, όχι μόνο ένας διεφθαρμένος υπάλληλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κριτήρια για τη διαφάνεια τέτοιων διεθνών δομών για να ξέρουμε, για να μπορούμε να ταυτίσουμε ευκολότερα ποιος ακριβώς είναι ο ένοχος. Αυτά θα τα πω πιο λεπτομερώς αργότερα, ιδιαίτερα για τους φραγμούς προς την ανάκτηση. Αυτό είναι το κύριο θέμα που μου ζητήθηκε να αναπτύξω σήμερα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόγραμμα που είχα αναλάβει που το ονομάσαμε Puppet Masters. Πώς δηλαδή θα διασφαλίσουν οι διάφορες χώρες ότι έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για όσους κρύβονται πίσω από επιχειρησιακές δίθεν δομές. Τώρα, αυτά διεθνώς, αλλά από την Αραβική Άνοιξη και μετά ιδίω πρέπει να γίνει προσπάθεια και αναχώρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ανάκτηση των κεκλεμένων περιουσιακών στοιχείων για να υπάρξει επιτυχής ανάκτηση. Αυτό καθίσταται όλο και σημαντικότερο τμήμα της δουλειά μας. Σας φαίνεται ίσως πεζό και απλό, αλλά είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που κάνουμε, δηλαδή πώς συνδυάζουμε τις δύο πλευρές, το, την υπηρεσία του ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα για να και είμαστε οι διαμεσολαβητές ας πούμε μεταξύ των θυμάτων και των δικαστών, των, των δικαστών. Και έρχομαι τώρα στο πρώτο πρόβλημα, στον πρώτο φραγμό προς τις ανακτήσεις που όπως σας είπα και πριν είναι το θέμα που έχω αναλάβει σήμερα. Ο μεγαλύτερος φραγμός για τις ανακτήσεις, το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει κάποια χώρα που ζητάει ανάκτηση είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Πριν από δύο χρόνια η Επίτροπος Ρέντινγκ έγραψε μία έκθεση που αναφέρει ακριβώς αυτό γιατί οι κατασχέσεις δεν γίνονται όπως πρέπει ιδίως διαμεθοριακά στην Ευρώπη γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών μιας χώρας και άλλης. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης υπάρχει ακόμη και μεταξύ σχετικά ομογενών, σχετικά παρόμοιων χωρών όπως μεταξύ της Ένωσης. Αυτό φάνηκε και από την Αραβική Άνοιξη. Ένας από τους ρόλους μας λοιπόν είναι να συνδυάσουμε τα μέρη για να συζητήσουν και να συνεννοηθούν, για να είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα του ενός και ποιο του άλλου. Μια χώρα της Αραβικής Άνοιξης ας πούμε μετά την Επανάσταση ζητάει ανάκτηση των εκατομμυρίων που έχουν κλαπεί πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η χώρα αυτή καταλαβαίνει και τους νομικούς φραγμούς και εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει και δυσκολίες. Η συνεννόηση λοιπόν των συμβαλωμένων σας έχω αναφέρει εδώ και ορισμένα ονόματα δικτύων, Κάριν, Αρίν, Σαστάρ, με την Ιντερπολ Συνδυασμός λοιπόν συνεννόηση των μερών. Άλλος γενικότερος φραγμός είναι η έλλειψη πόρων. χρηματικών, ανθρώπινων πόρων και γνώσης. Άρα και capacity building για να μπορέσουν οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τους δημοσιονομικούς ελέγχους και να υπάρξει αμοιβαία νομική βοήθεια. Και σχετικό με αυτό, άλλος φραγμός, η έλλειψη μιας γενικότερης παγκόσμιας πολιτικής για τις ανακτήσεις, στρατηγική και συντονισμός, ιδίως λόγω πολιτικών πιέσεων, σε χώρες όπου έχει μόλις πέσει κάποια διεφθαρμένη κλίκα πρέπει να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη στρατηγική τα επόμενα βήματα. Οι πολιτικοί ζητούν άμεση δράση συνήθως, αλλά πρέπει πριν εφαρμοστεί η δράση να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν τις σωστές προτεραιότητες, ότι δεν στέλνουν 150 αιτήσει ανάκτησης ταυτόχρονα, αλλά στοχεύουν τα πράγματα και έχουν κάποια στρατηγική άποψη. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να υποβοηθήσουμε χώριους μηχανισμούς συνεννόησης, να υπάρχει ένας υπεύθυνο ή μία υπηρεσία υπεύθυνη για την ανάκτηση, οι άλλες χώρες να γνωρίζουν ότι αυτή η υπηρεσία ασχολείται με το θέμα και να δημιουργηθούν ειδικέ μονάδες έρευνας που να ασχοληθούν με αυτό. Τώρα μερικά από τα νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Χάρηκα που ο προηγούμενος ομιλητής ανέφερε το θέμα του ότι δεν υπάρχει κανένας ενιαίος μηχανισμός επιβολής όλων αυτών. Όταν διώκεται κάποιος για διαφθορά μπορεί να υπάρχουν ασυλίες, μπορεί να, να είναι ο κατηγορούμενος να έχει υπερβολικά μεγάλη εξουσία και να προστατεύεται. Πολλοί λόγοι μπορεί να υπάρξουν για την παρεμπόδιση για να μην μπορέσει κανείς να καταδικάσει τον κύριο υπεύθυνο. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να γίνει η ανάκτηση. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα αυτό κάνει ακριβώς, ε, κέρδη αποφέρει και μπορούν πάντοτε να παγώσουν ή να ανακτηθούν τα κέρδη αυτά, ακόμη και αν δεν καταδικαστεί ο υπεύθυνο. Άλλο θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά είναι ότι δεν υπάρχει ένας γρήγορος μηχανισμός παγώματος των κερδών ή των περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων. Πρέπει να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός για το πάγωμα, γιατί η κατάσχεση είναι κάτι που κρατάει πολύ χρόνο. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας άμεσος μηχανισμός παγώματος τουλάχιστον. Και αυτό πολύ σημαντικό νομικά. Αν θέλουμε να καταλήξουμε στην ανάκτηση. Μπορεί να γίνει δικαστικά και να εφαρμοστεί με φάνταστο τρόπο, με καταλόγους κυρώσεων για το πάγωμα του λογαριασμού ας πούμε κάποιου. Είναι πολύ καλός τρόπος για να αρχίσει η διαδικασία της ανάκτησης. Και τέλος, είναι το θέμα που ότι σε μερικές χώρες αν θέλει κανείς να έχει πληροφορίες για το λογαριασμό κάποιου μπορεί να τους απαντηθεί μόνο με την άδεια του ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν σημαντικό και οι χώρες να μην αντιδρούν έτσι να μην δηλαδή προειδοποιούν τον υπεύθυνο ότι θα του γίνει έρευνα. Δεν ξέρω αν επικαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Αυτά είναι νομικοί φραγμή που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, λειτουργικοί φραγμή. Δεν υπάρχουν κατάλληλα ή σαφή σημεία επαφής μεταξύ των χωρών που ζητούν ανάκτηση. Οι περισσότερες έχουν περάσει από πολιτική ταραχή και δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την έρευνα ο εισαγγελέα, το Υπουργείο Εσωτερικών ή άλλο. Ενώ οι άλλες χώρες θέλουν να ξέρουν ποιος είναι ο υπεύθυνος της έρευνας και σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν. Και σε αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε. για να υπάρχει, να διασφαλίζεται χώριο συντονισμός και να βοηθηθούν έτσι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα να συνεννοηθούν. Και αυτό ακούγεται πεζό, αλλά είναι πολύ πραγματικό και πολύ συχνό. Η φορμαλιστική προσέγγιση τώρα είναι ένας άλλος φραγμός. Πολλές χώρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν νόμους που προβλέπουν ότι αν το εισόδημά σας είναι μερικές χιλιάδες το μήνα ενώ έχετε περιουσία εκατομμυρίων, αυτό μπορεί να είναι τεκμήριο. Και θα αρκούσε για να μπορέσετε να κατηγορηθείτε για παράνομο πλουτισμό. Αλλά δεν το δέχονται αυτό όλες οι χώρες αν υπήρχε γενικώ το κριτήριο του τεκμηρίου του πλουτισμού, θα διευκολύνονταν τα πράγματα. Αν ερευνήσει κανείς τα πράγματα θα δει ότι συνήθως αυτός ο περίεργος πλουτισμός οφείλεται σε παράνομη δραστηριότητα. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να αντιδράσει κανείς ακόμη και αν δεν υπάρχει ο σχετικός νόμος σε κάποια χώρα το τεκμήριο του πλουτισμού δηλαδή. Όποιο και να είναι το όνομα της ε, αντίδρασης που θα δώσουμε, που θα αναλάβουμε, μπορούμε να ερευνήσουμε. Να ενθαρρύνουμε τις χώρες να μην είναι πολύ φορμαλιστικές αυτά τα κριτήρια, η τεκμήρια, η απουσία τους. Και κάτι άλλο, πολλές από τις χώρες αυτές για πρώτη φορά αναλαμβάνουν έρευνα για ανάκτηση. και δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς πρέπει να το κάνουν επειδή δεν έχουν τέτοια ανάλογη εμπειρία. Ούτε οι εισαγγελείς, ούτε οι ερευνητέ γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Και μπορεί οι πρώτες τους προσπάθειες να είναι ατελείς, να μην συμφωνούν πλήρως με τα απαραίτητα νομικά κριτήρια και, γι αυτό, και σε αυτό τις βοηθάμε. για να υποβάλουν τις αιτήσει τους όπως πρέπει. Και στα διεθνή πιστοτικά κέντρα προσπαθούμε να πούμε ότι πρέπει να βοηθήσουν την ετούσα χώρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος, δύο άλλοι φραγμοί. Η δυνατότητα ή μη να ταυτίσει μια χώρα λογαριασμού σε άλλη πολιτών της βέβαια. Δεν υπάρχουν τέτοια διεθνή μητρώα και εμεί ζητάμε την εφαρμογή τους, την έγκριση τους, να ξέρει μια χώρα αν οι πολίτες της και ποιοι έχουν ξένους λογαριασμούς. Η Ευρώπη εδώ πρωτοπορεί και εμείς προσπαθούμε να υπάρχει ένας μηχανισμός με τον οποίο να μπορεί μια χώρα πολύ σύντομα να δει από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς αν υπάρχουν λογαριασμοί πολιτών της, συγκεκριμένων πολιτών της. Τέλος, κάτι για το οποίο θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες ολόκληρες, είναι ότι δεν έχουμε συνήθως ποτέ στοιχεία για την ιδιοκτησία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Φυσικά ο εγκληματίας δεν βάζει στο δικό του όνομα τα περιουσιακά του στοιχεία. Συνήθως κάποια διεθνούς εταιρεία είναι τυπικά τα περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να έχουμε όμως πληροφόρηση για να γνωρίζουμε ανήκει, σε ποιον ανήκει τι. Ποιος ελέγχει μια εταιρεία. Υπάρχει αυτό το βιβλίο The Puppet Masters που σας είπα πριν, η καραγκιοζοπέκτε, για να, όπου που γίνονται προτάσεις για μέτρα όπως η βελτίωση της πληροφόρησης για τα επιχειρησιακά μητρώα και υπάρχει η αναγκαιότητα οι τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να χορηγούν αυτές τις πληροφορίες, πράγμα που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Πολλές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν δίνουν τέτοιες πληροφορίες. Επίσης, οι λογιστές και δικηγόροι που λειτουργούν σε αυτές τις διεθνείς εταιρείες πρέπει και αυτοί να διαθέτουν όλες τις πληροφορίες, να μην λένε εγώ είμαι ουδέτερος ε, προμηθευτής ε, υπηρεσιών. Όχι, πρέπει να ξέρει τα πάντα αυτός που αναλαμβάνει τέτοια δουλειά. Θα μπορούσα να σας δείξω πολλά περισσότερα, πολλές περισσότερες διαφάνειες, αλλά σας ευχαριστώ εδώ. Σταματάω εδώ. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω στους ε, να πάρα πολύ αυτό που είπε ο κύριος Μασερδίτσι. Δηλαδή, εμείς εκφράσαμε την ανησυχία μας ε, για μια σειρά από θέματα τα οποία λείπουν, λείπουν παντελώς από την οδηγία περί κατασχέσεων σχετικά με την ε, επαναχρησιμοποίηση των κατασχεθέντων αγαθών. Θέλω λοιπόν τώρα να δεχτούμε τις ε, ερωτήσεις ε, που θα απευθύνεται στον κύριο Μασερβίζη, ο οποίος ε, πρέπει να εξαφανιστεί μετά ταχύτατα, γιατί συμμετέχει σε μια τριμερή συνάντηση. Παρακαλώ να είσαστε σαφείς δυνατόν. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία ότι το ποινικό, το εγκληματικό σύστημα, το εγκληματικό σύστημα οδηγεί στο ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, στις αστυνομικές δυνάμεις και στη δικαστική εξουσία. Να υπάρχει κάποια ευελιξία. Το είπατε εσείς ότι θα πρέπει το εγκληματικό σύστημα να το χτυπήσουμε στην καρδιά. Και έτσι λοιπόν ε, χρειαζόμαστε και ένα αποτελεσματικό σύστημα για να ανακτήσουμε τα αγαθά από τη μαφία και να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Ακόμα και για ε, συμβολικές αξίες είναι σημαντικό οι αξίες αυτές να χρησιμοποιούνται για την κοινωνία. Αναφερθήκατε σε σκέψεις ε, που κάνετε και με πείσατε πλήρως, αλλά από την ακρόαση που είχαμε και στη Ρώμη ε, διεφάνει ότι ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τα αγαθά ανακτηθέντα από τη μαφία είναι ότι αυτά είναι αντικείμενο βανδαλισμού, είναι πολλές φορές υποθηκευμένα αγαθά και εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Εσείς λοιπόν μας είπατε ότι δεν υπάρχει η νομική βάση έτσι ώστε η οδηγία αυτή να διαχωρίζεται πλήρως από ε, τα αγαθά τα οποία κατάσχονται από τη μαφία. Μας είπατε επίσης και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχουν οι διατάξει εκείνε ε, στα κράτη-μέλη που να επιτρέπουν και τη χρήση διαφορετική εμπειρία. Αυτό συμβαίνει κυρίω ε, στην Ισπανία. Βεβαίως ε, αυτό είναι ο στόχος της ε, εναρμόνισης των ε, νομοθεσιών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ένα μοντέλο αναφορά το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα άλλα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μας λοιπόν είναι καθοριστική σημασία να υπάρχει κάτι τέτοιο ε, και λόγω του ότι ένα αγαθό που αφαιρείται από τη μαφία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε για συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι λοιπόν θα ήταν ευκταίο μέσα από μια διάταξη, αν υπήρχε κάποια διάταξη, να εξετάσει κανείς ουσιαστικά το θέμα αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι ακόμα πιο σαφής. Ο ε, διευθυντής μας είπα προηγουμένως πράγματι αυτό λείπει στο νέο πακέτο, αλλά θέλω επίσης να σας πω ότι ε, υπάρχει πρόβλημα ε, και το όλο αυτό πακέτο να νοθευτεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον διευθυντή να μας πει τι μπορεί να κάνει η διεύθυνσή του έτσι ώστε έστω και αυτά τα λίγα που υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν σωστά, να μην υπάρχει κίνδυνος ε, νόθεψης ε, και πολύ ήπιας ε, διαμόρφωσης, γιατί τελικά θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο δεν θα είναι καθόλου χρήσιμο. Γιατί δεν θα υπάρχει η εναρμόνιση των νομοθεσιών. Ορισμένα κράτη είναι ακόμα επιφυλακτικά και βρίσκονται στην άμυνα περισσότερο παρά στην επίθεση. Η κυρία Βάιλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να αναφερθώ λιγάκι στο σχέδιο οδηγίας του Μαρτίου. Ε, είπατε δηλαδή ότι λόγω της ε, νομικής κατάστασης ε, με βάση το άρθρο 83 δεν μπορείτε να καταθέσετε πιο προχωρημένες προτάσεις. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση όταν δηλαδή συνενέσουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να κατατεθούν προτάσεις ε, Παραδείγματο χάνει για την ένταξη σε αυτά τα τοπικά ε, προγράμματα ε, τα οποία σε ορισμένα κράτη-μέλη αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα. Αυτό που με εκπλήσει είναι που λέτε ότι η οδηγία μπορεί να νοθευθεί. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από πλευρά του Κοινοβουλίου αλλά από το Συμβούλιο που έχει κάπως αφήσει να νοηθεί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο. Εδώ όμως το Κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί στεναρά. Αν δηλαδή συμφωνήσει η Επιτροπή Λίμπε ε, και η Επιτροπή δική μας εδώ, η ΚΡΙΜ, να κατατεθούν οι σχετικές ε, τροπολογίες και έτσι θα εκπέμψουμε χειρό μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι δηλαδή εμεί θέλουμε κάτι να γίνει και ότι αυτή η ασάφεια στην νομική βάση θα πρέπει να αρθεί. Το κάναμε και στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Βέβαια πρέπει να ονοματίσουμε στην περίπτωση αυτή τα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούν να παραμένουν έτσι χαλαρά και αδέσμευτα. Και θα με ενδιαφέρει, α πούμε, αν αυτό αφορά τη δική μου την πατρίδα, τη Γερμανία ή ποιε χώρες, μήπω τους Βρετανούς ή κάποιου άλλους, οι οποίοι δεν επιθυμούν να υπάρχει εναρμόνιση των νομοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι εισηγητές αυτή την ακρόση, αλλά και κατά τους ε, τελευταίους μήνες μας είπαν ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί, μεγαλύτερη εναρμόνιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο στην πατρίδα τους, αλλά ε, να συμπεριλάβουν στο δίκαιό τους ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι έχει αποδειχθεί ε, σωστό. Έχετε λοιπόν τη δική μας την υποστήριξη. Δεν άκουσα κανένα που να τάσετε υπέρ μιας, ε, ενός πιο ισχυρού ευρωπαϊκού κανονισμού. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε στις ε, πατρίδες μας, έτσι όπως είπε και ο εκπρόσωπος Κομισιόν, να μην υπάρξει η νόθευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κυρία Μπορσελίνο και εγώ έχουμε προτείνει μία τροπολογία για το 83-2. Έλεγα ότι με τη συνάδελφο Μπορσελίνα είχαμε προτείνει ως νομική βάση το 83.2 της συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή ε, το θέμα αυτό ε, πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η κυρία Ματιού. Ευχαριστώ. εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη γνώμη της συναδέλφου, αλλά είμαστε στην Επιτροπή Κρίμη, θα πρέπει να πάμε στη ΛΥΜΠΕ. Νομίζω ότι και συνάδελφος ε, το καταλαβαίνει ότι εδώ ε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ πραγματικά απογοητεύτηκα με τη συζήτηση στη ΛΥΜΠΕ και να σας πω την αλήθεια έχουμε συναδέλφους ε, που περιχαρακώνονται πίσω από το κράτος μέλος τους ε, και που βάζουν φρένο στη διαδικασία. Και είναι κρίμα, κυρίως ό,τι αφορά τη Γαλλία. Δεν ε, υπάρχει βουλή συναρμόνησης. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ναι, και θέμα πλειοψηφίας και υπό την προηγούμενη κυβέρνηση νομίζω το ίδιο θα ισχύει και είναι κρίμα γιατί δεν υπάρχει βούληση να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα και σε αυτή την οδηγία. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως ε, να λειτουργήσουμε ως εξής. Ε, ίσως θα έπρεπε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση αυτή να μην ασχοληθούν τόσο πολύ με το τι σκέφτεται η κυβέρνησή τους. Και ίσως ε, αυτό είναι ένα βήμα ε, που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει οι συνάδελφοι που παρευρίσκονται εδώ και συμμετέχουν στην Κρίνη να συνεδριάσουν και να συζητήσουν με τους συναδέλφους από τη Λίβη και να τους πούνε ότι εμείς είμαστε υπέρ αυτής της γιατί είναι ο μόνο τρόπος να καταπολεμήσουμε τη μαφία και θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό στις αντίστοιχες ομάδες μας και να πείσουμε τους συναδέλφους γιατί αυτή είναι η δυσκολία σε κάθε πολιτική ομάδα. Αν ε, θέλουμε να προχωρήσουμε, μπορούμε και νομίζω ότι υπάρχει πραγματικό μπρεντεφέρ μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Θα είναι ιδιαίτερα πολιτική συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Τα βάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τις προηγούμενες επεμβάσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η ειδική επιτροπή που έχει προσωρινό χαρακτήρα να βρει μια πολύ σαφή στρατηγική προκειμένου να συμμετέχει και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, σε αυτό το εγχείρημα. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει τη σχετική έκθεση Μακοβέη. Θα έπρεπε να συνεδριάσουμε από κοινού με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά και με την ε, Επιτροπή για τους Προπολογισμούς και την Επιτροπή Αναφορών. Γιατί και εδώ κάνω μια άμεση ερώτηση στον κύριο Ματσερβίση για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα της νομικής βάσης ε, για να δημιουργήσουμε αυτό το ταμείο με τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που θα μπορούσε να δώσει ε, πολιτική προβολή στην κατάσχεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα ήταν να δημιουργηθεί ένα ταμείο στο οποίο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες με ένα σύστημα παρόμοιο με τα πιλωτικά σχέδια που χρησιμοποίησαμε στην Επιτροπή Προπολογισμού ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι λοιπόν θα είχαμε και κοινοβουλευτικό έλεγχο και δημοκρατικό και πολιτικό έλεγχο αλλά όμως οι πολίτες, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, των, πληγέ, των πληγισών περιοχών θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια και αυτό να γίνει μέσω της Επιτροπής Αναφορών. Έτσι λοιπόν θα κατορθώναμε να μπλέξουμε τέσσερις επιτροπές, από τις οποίες οι δύο είναι πολύ ισχυρέ σε αυτό το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών μάλιστα πρέπει να βρει και το αντικείμενό της για να μπορέσει να κερδίσει σε πολιτική σημασία. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι την πλευρά του Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να έχουμε την κατάλληλη πλειοψηφία για να προωθήσουμε αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη. Λοιπόν, αυτό για το πρώτο θέμα. Τώρα, θα είμαι πολύ γρήγορο γιατί έχω και άλλε ερωτήσει. Ε, ο κύριο από την Παγκόσμια Τράπεζα μίλησε για θέματα αμοιβέ εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και άλλων περιοχών του πλανήτη. Εγώ βλέπω εδώ μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ των πληροφοριών ε, που, που δίνουμε στο πλαίσιο της ε, SWIFT και FTP από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για λόγους καταπολέμησης τρομοκρατίας ή διασυνοριακού εγκλήματος και κατόπιν των πληροφοριών που εμείς δεν αποκτούμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και το οικονομικό έγκλημα, το οποίο είναι και αυτό διασυνοριακό έγκλημα. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ματσερβίση, μέχρι ποιο σημείο εμείς μπορούμε στην αναθεώρηση της εφαρμογής της TFTP να ζητήσουμε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πληροφορίες για τους ε, τελικούς δικαιούχους ε, των τραπεζικών λογαριασμών ε, και των ακινήτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και καθώς μιλάμε για τραπεζική ένωση θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και το θέμα του καθολικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών. Και νομίζω ότι πρέπει να επιμείνει το Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπιλνιούτον Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσε και δύο παρουσιάσει. ευχαριστώ. Κανεί δεν κοιμόταν. Ε, εδώ και αναφέρθηκατε στους φορολογικούς ε, παραδείσους ε, και δυστυχώς υπάρχουν χορηγία από ορισμένα κράτη-μέλη και δυστυχώς και από το δικό μου κρατη μέλη. Αν δεν μπορούμε να εξελίψουμε τους φορολογικούς παραδείσους, τότε υπάρχουν συνεχώς ανοιχτά παραθυράκια για τους κακούς. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους φορολογικούς παραδείσους και για τον κύριο Μασερβίση. Ξέρουμε όλοι ότι τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται να συνεργαστούν, το ίδιο ισχύει για κάθε τομέα ευρωπαϊκής δραστηριότητας. Να προτείνω αυτή η επιτροπή και η έκθεση του κ. Λεκολίνου, που θα παρουσιαστεί τον επόμενο χρόνο, είναι μια πραγματική ευκαιρία για να ξεπεράσουμε τι αντιρρήσει των κρατών μελών. Γιατί αν Κομισιόν και το Κοινοβούλιο συνεργαστούν λέγοντα, α δούμε το μέγεθο του κλίμακα αυτού του προβλήματος, επί το οποίο εργαζόμαστε για χρόνια», η συνολική απολύτω εισοδήματο από τα κράτη-μέλη και συνολική απώλεια θέσεων εργασία είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Και να απευθύνουμε έκκληση στο κοινό και έχουμε τον ε, κύριο Γιακολίνο, την κυρία Αλφάνο, εσά τον Επίτροπο που όλοι λέτε αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε του πολίτε και να πούνε πολίτε στις εθνικέ κυβερνήσει μα, σας παρακαλούμε έλεος, κάντε κάτι. Έχουμε μια ευκαιρία να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Επομένω, αν η Κομισιόν μπορεί να μα βοηθήσει με όλα τα αριθμητικά στοιχεία και τι λεπτομέρειε που θέλουμε για να ε, παρουσιάσουμε πλήρως αυτή την υπόθεση στο κοινό, έχουμε μια ευκαιρία. Αυτή είναι μια πρόταση για τον άλλο κύριο που έχει τόσο πολύπλοκο όνομα αλλά πολύ καλή προφορά Βιάζεται ο διευθυντή, επομένω ε, μόνο τι ερωτήσει για τον κύριο Μεσερβίση δεν ρωτή, μπορώ να ρωτήσω τώρα, δηλαδή τον ε, άλλο μιλητή. Όχι, όχι, σε λίγο. Ευχαριστώ, Μπιλ. Η κυρία Γιαννάκου τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, τα ίδια ερωτηματικά που ετέθησαν για την οδηγία έχω και εγώ. Ε, έχω την εντύπωση όμως ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση το Συμβούλιο. Όντως δεν υπάρχει σωστή συνεργασία και όχι μόνο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ε, η διαφθορά που παράγεται όταν νόμιμες επιχειρήσεις για να πάρουν προμήθειες του δημοσίου στις χώρες της Ευρώπης χρηματοδοτούν υπαλλήλους, πολιτικούς και άλλους. Και έχουμε τέτοια περιστατικά για υποθέσεις διαφθοράς όπου βέβαια στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία έκλεισαν τους φακέλους με πολιτικά κριτήρια. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη εφαρμογή για όλους. Ούτε το δικαστικό σύστημα συνεργάζεται και πρέπει να σας πω ότι στις υποθέσεις κατασχέσεως περιουσιών έχουμε το εξή φαινόμενο, παραδείγματο χάρη στη χώρα μου. Παγώνουν οι λογαριασμοί των υπόπτων, οι ύποπτοι διαφεύγουν στο εξωτερικό Υφίσταται η οικογένειά τους τις συνέπειες του παγώματος και εν συνεχεία κάποια στιγμή ξεπαγώνουν οι λογαριασμοί, ο φυγόδικος έχει εξαφανιστεί και δεν εφαρμόζεται η δικαιοσύνη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε και επίσης ένα σχόλιο που θέλω να κάνω. Στη χώρα μου είναι πολύ αυστηρές ποινές για όλα. Καταλήγουν όμως στο τέλος στην ατιμορρησία. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις τέτοιες που πρώτον να μην μπορεί κανείς να διαφύγει σε άλλη χώρα όπου υπάρχουν ευνοϊκότερες συνθήκες. Πρέπει δηλαδή το σύστημα να είναι ενιαίο. Και δεύτερον πρέπει το σύστημα να είναι ισορροπημένο ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται αυτά που προβλέπει και όχι να υπάρχουν παράθυρα διαφυγής. Αυτά είναι τα δύο σημεία που έχουμε από την εμπειρία μας σε τέτοιες υποθέσεις που όντως είναι πολύ δύσκολες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία παρέμβαση ο κύριος Τάι. Η κυρία Τάι. Εγώ θέλω να κάνω τον δεύτερο μιλητή. Αν θέλετε, μπορώ να τι κάνω αργότερα. Πολύ ωραία. Δίνουμε λοιπόν ε, το λόγο στον ε, Διευθυντή Μανσερβίζη για να απαντήσει. Σα ζητώ συγγνώμη αλλά έχω μία συνάντηση για το ασύλο, έτσι λοιπόν ε, πρέπει να βιαστώ και να τα καταφέρω κάπως. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρατηρήσεις, ε, οι οποίες ήταν επικριτικές, αλλά ακολουθούν και τη σωστή κατεύθυνση για να πετύχουμε το μέγιστο. Να πω λοιπόν πρώτα απ' όλα το εξής. Ε όσον αφορά το ρόλο αυτή τη επιτροπή, Εντάξει, δεν είναι δική μου δουλειά να το καθορίσω αυτό, αλλά αυτό που φοβάμαι είναι ότι αν οι διαπραγματεύσεις ε, καθοδηγούνται από την συνηθισμένη λογική, δηλαδή να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό λαμβάνοντας υπόψη ακαμψίες και αγκυλώσεις και αν δεν γίνει απολύτως κατανοητό ότι αυτό ναι μεν είναι ένα νομικό εργαλείο όπως όλα τα άλλα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια, ε, υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση του οργανωμένου εγκλήματος, άρα δηλαδή πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες. Αν δεν τα κατανοήσουμε όλα αυτά, εντάξει θα καταλήξουμε σε ένα συμβασμό, ο οποίος όμως θα είναι μόνο στα χαρτιά και όχι στην ουσία. Βεβαίως εναπόκειται σε εσά να αποφασίσετε, αλλά αυτά που είπατε κύριε Νιούτον Ντάν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ουσιαστικό να ε, καταδείξουμε αυτά που σας είπα με στοιχεία, με εκστρατείες και βεβαίως ε, ε, και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι καθοριστική. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η πρότασή σας ε, θα είναι πολύ χρήσιμη και στην Επιτροπή Λίμπε και αλλού. Σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο ένα συμβασμό στα χαρτιά, δεν είναι αυτός ο στόχος ή θα τα ε, καταφέρουμε καλύτερα ή θα χάσουμε μία ευκαιρία. Θέλω να υπογραμμίσω, όπως είπε ακούστηκε και στο τέλος, ότι αν τελικά δεν έχουμε ένα ενιαίο καθεστώς το οποίο να επιτρέπει να δεσμεύονται αγαθά, να μην υπάρχουν παραθυράκια, ακόμα έστω και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτές όμως, έστω και αυτές, το 80% αυτών αφορά προσπάθειες του οργανωμένου εγκλήματος για να συγκαλύψει, να κρύψει τα κέρδη από παράνομες πράξεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν ισχυροί νόμοι σε εθνικό επίπεδο που εφαρμόζονται. Το θέμα των φορολογικών παραδείσων είναι σημαντικό. Αλλά θα θυμάστε όταν συζητάγαμε την οδηγία για την φορολογία εσόδων, πράγματι Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ε, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για μας είναι η πρόφαση να μην κάνουμε τίποτα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο αναδυόμενος κόσμος και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχουν διμερεί συμφωνίε, πιο αποτελεσματική συνεργασία με τις ε, τρίτες χώρες, αλλά όπως δείχνουν τα στοιχεία, ε, το πιο σημαντικό είναι η δική μας η κοινή αγορά. Αν λοιπόν ε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα κατά, τότε δεν είμαστε αξιόπιστοι Άρα δηλαδή είναι δεσμευτικό να εναρμονίσουμε την προσέγγιση μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκε προηγουμένως ότι θα πρέπει ε, να αναφερόμεθα και εμείς ε, στο FTP που καλύπτει ε, σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Αλλά όμως σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται από τις ΗΠΑ. Αρχίζουμε τώρα λοιπόν να καλύπτουμε ότι πολλά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν και αυτά τις ε, πληροφορίες για δικούς τους ίδιους σκοπούς. Ας το δούμε λοιπόν αυτό ε, με κάποιο πιο αυστηρό τρόπο και ας προτείνουμε κάποιες δράσεις. Αν λοιπόν το θέμα δεν γίνει κατανοητό, πράγματι ε, θα παραμείνει κατακαιρματισμένο. Κάτι άλλο που αφορά ε, τα κονδύλια, τα χρήματα. Άκουσα τις διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν και εγώ με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές. Ξέρετε τις διαπραγματεύσεις ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς ε, τρέχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και ξέρετε ότι το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ε, οδήγησε και σε τίποτα το σημαντικό. Εντάξει, το να υπάρξει δική γραμμή στον προβλησμό, καλό θα ήταν αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Ανταυτού, αυτό που προτείνουμε εμείς, ένα ταμείο εσωτερικής ασφάλειας, που θα είναι πιο ευέλικτο, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει, ε, αν θέλετε, πιλωτικά προγράμματα. Αυτή είναι μια ιδέα που βεβαίως εξαρτάται από το τελικό αποτέλεσμα και τη νομική βάση που θα εγκριθεί. Άρα δηλαδή και εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί έχοντας ε, κατά νου το τι μπορεί τελικά να προκύψει. Και βέβαια και τα ποσά παίζουν ρόλο. Γιατί αν τελικά αποφασιστεί ότι το 70% των κονδυλίων ε, θα το διαχειρίζονται, θα υπά, για αυτά θα υπάρχει κοινή διαχείριση, αυτό θα δυσχεραίνει την κατάσταση. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ε, ο στόχος είναι να υπάρχει κάτι εφικτό. Όσον αφορά τη νομική βάση, νομίζω απάντησα. Το άρθρο 83 είναι το μόνο κατάλληλο. Μιλάμε λοιπόν για εναρμόνιση με βάση νομοθεσία που ήδη υπάρχει. Ε, όμως είναι σχετικά μόνο αποτελεσματική. Δεν είναι εναρμόνιση, αλλά μάλλον συνεργασίας μεταξύ ιδιοκτικών αρχών αν δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό νομικά, ας το κάνουμε με τα συνοδευτικά μέτρα όπως τις κατασχέσεις με κοινωνική χρήση των περιουσιακών στοιχείων. Όσο για την Πασαρέλα, ένα θεωρητικά ναι, αλλά αυτό απαιτεί ομοφωνία. Κι αν υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν όλα αυτά, τότε καλύτερα να εφαρμόσουμε μέτρα που να απαιτούν μόνο ενισχυμένη πλειοψηφία στη συναπόφαση. Γιατί εδώ δεν αποζητούμε συμβιβασμό αλλά λύση. Διότι όλοι μας κάποτε θα χρειαστεί να κάνουμε επιλογές και να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε για τι πράγμα μιλάμε. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που φεύγω, αλλά έχω εδώ ένα συνεργάτη που μπορεί να απαντήσει σε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, ξαναξεκινάμε τη συζήτηση. Ε, ερωτήσεις προς τον κύριο, ε, από την κυρία Μακιντάιρ. Προς τον κύριο Βαντερντές. Ε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Δεν άκουσα την ε, πρώτη παρουσίαση, αλλά άκουσα τη δικιά σας. Και κατάλαβα ότι είναι σημαντικό να καταζητήσουμε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Πολλές φορέ όμως άκουσα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η ε, σωστή δίωξη. Και έγραψε, τώρα έγραψε μάλιστα, είπατε ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πολύ ισχυροί για να ε, υποστούν τη δίωξη. Αυτό όμως για μένα είναι φοβερό. Με, με τρόμαξε η δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει παντού σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως επίσης και το κράτος δικαίου. Παντελώς απαράδεκτο το να λέγεται ότι μερικοί είναι πολύ ισχυροί για να διωχθούν. Απλά ήθελα έτσι να εκφράσω τον τρόμο που με κατέκλυσε. Κατά τα άλλα, ε, σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε, στο πρωτόκολλο 36 το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεται ως μια χώρα που μπορεί να αυτοεξαιρείται από μέτρα εσωτερικής ε, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Ποια από τα υπάρχοντα μέτρα, τα κείμενα μέτρα, εάν αποσύροντο θα οδηγούσαν σε επιδείνωση της κατάστασης και θα επέφεραν και περισσότερους φραγμούς, όπως εσείς τους εξηγήσατε. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα υπάρξουν και άλλα εμπόδια και ποια. Και υπάρχουν μήπως ε, κάποιοι τομείς ε, που σας απασχολούν ιδιαίτερα. Πολύ ωραία. Ο κύριος ε, Νιούτον Μπιλ, έχει το λόγο. Ορίστε Μπίλ μου. Μπίλ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Απαντούσα στην κυρία τα ότι ένα ε, παράδειγμα ανθρώπου με πολύ, που είναι πολύ ισχυρό για να διωχθεί ήταν ο κύριος Μπερλουσκόνη. Τέλο πάντων. Ευχαριστώ. Θαύμασα το, τα αγγλικά του ομιλητή με το βελγικό όνομα. Τα, η φορολογική παράδειση είναι ένα θέμα, αλλά ανέφερε επίσης και το ενδιαφέρον θέμα του παράνομου πλουτισμού δηλαδή χαμηλά έσοδα, από μεγάλη περιουσία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν τεράστια σπίτια και κτήματα με πολύ χαμηλό μηνιαίο εισόδημα. Μπορεί να οφείλονταν και αυτά αρχικά σε εγκληματική δραστηριότητα, αλλά είναι των αριστοκρατών, ξέρετε. Έπειτα μιλήσατε για τους καραγκιοζοπέκτα στο βιβλίο Puppet Masters. Έχετε κανένα αντίτυπο. Έψαξα στο Google και λέει ότι είναι κινηματογραφικό έργο στο οποίο ορισμένοι εξωγήινοι έρχονται ως άνθρωποι. Είναι τόσο ενδιαφέρον και το βιβλίο σας. Αν έχετε αντίτυπα παρακαλώ να μας δώσετε. Ο κύριος Γιακολίνος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τους φορολογικούς παραδείσους, αναφέρθηκε ο κύριος Νιούτον Ντάν τώρα για το θέμα των τραπεζών, για το ρόλο των τραπεζών. Αν θα μπορούσε να χρήσιμη μια τραπεζική ένωση για πιο αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των ζητημάτων. Δηλαδή, αν υπάρχει μια διατραπεζική διακυβέρνηση στα πλαίσια της ε, τραπεζικής ε, Ένωσης, αν θα ήταν κάτι χρήσιμο. Επίσης, ε, ποιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, η δέσμευση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να έχουμε μεγάλη ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης. Χρειάζεται και μεγάλη ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ε, και δεν υπάρχει πάντοτε, γιατί ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να είναι ε, το αλάτι αυτό των συνδέσεων συχνά λείπει. Ε, αναφέρθηκε κάποιος στον Καντάφη. Θυμόμαστε τις αντιδράσεις τότε. Δεν είναι όλοι ο Καντάφη, αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ε, οι οποίες εκδηλώνονται σε κάποιες περιπτώσεις. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η οδηγία για την ε, καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων και τι θεωρείται από τις αξιολογήσεις για το θέμα της δέσμευσης που συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και υπήρξαν για κάποιες άλλες εκθέσεις, γιατί πρόκειται για συμπληρωματικά μέσα και για την καταπολέμηση της νομοποίηση παράνομων εισόδων. όταν μιλήσατε για φορολογικού παραδείσου, μιλήσατε και για άλλα θέματα, αλλά στην Ευρώπη, χωρίς να δακτυλοδείξουμε, υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία είναι πάρα πολύ ανεκτικά και διαθέσιμα να δώσουν πληροφορίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από ε, κάποιο που το αξίζει. Βάσει της εμπειρίας σας, μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι να αναφέρουμε και τα ονόματα αν ε, ο μιλητής διαθέτει αυτά τα στοιχεία. Ο κ. Κύρκο, ευχαριστώ. Μιλώντας ως νομικός και ως κάποιος που έχει ξοδέψει πολλά χρόνια από την καριέρα του στην υπεράσπιση, στο δικαστήριο, Βλέπω ε, τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ε, ε, σε σχέση με το αν διώκονται ή όχι από τη δικαιοσύνη, αρκετά ενδιαφέρουσες και άκουσα ότι είπε και ο κύριος Νιούτον Ντάν, ο οποίος ε, αναφέρθηκε σε μια δίκη πολιτικού στην Ιταλία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα η υπόθεση του κύριου Μπερλουσκόνη και δεν θέλω να παρέμβω στα ιστορικά της Ιταλίας, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε πάρα πολλές χώρες είναι η πολιτική φύση του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών της εισαγγελία. Και αυτό με ανησυχεί πολύ. πολύ. Νομίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρητικά τουλάχιστον, ε, η εισαγγελία υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Θα πάρει μια απόφαση σε σχέση με αν υπάρχει μια πιθανή ε, καταδίκη, μια δυνατότητα καταδίκης ε, πριν προχωρήσει και αυτό πρέπει να το κάνει χωρίς καμία πολιτική πίεση από καμία πλευρά. Σε άλλες χώρες, να δούμε την Γαλλία, <laughs> όπου έχουμε μια εισαγγελία ε, συγκεκριμένη και το θέμα είναι ποιο διορίζει ποιον. Όποιο ε, διορίζεται απευθεία από πολιτικού φυσικά ε, μπορεί να υποστεί πολιτική πίεση. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να ζητήσουμε εδώ και αυτή είναι ενδιαφέρουσα ένδειξη και στι Ηνωμένε Πολιτείε γιατί πολλέ δουλειέ στην εισαγγελία είναι πολιτικού χαρακτήρα. Και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε τη δουλειά που κάνουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη επιτροπή για να δούμε πώς ε, θα μπορούσαμε να επιφέρουμε αποδοχή και κατανόηση στα κρατημέλη ότι η εισαγγελία θα πρέπει να είναι μη πολιτικού χαρακτήρα στο μέτρο του δυνατού. Θα έλεγα ε, σε ορισμένε περιπτώσει ε, είναι αδύνατο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο που επιδιώκουμε εδώ. Γιατί έχω δει πολλέ υποθέσει και η υπόθεση του κ. Παγκλουσκόνη αναφέρθηκε. Νομίζω ότι ο Μπίλ θα συμφωνούσε μαζί μου ότι δεν μιλούσαμε ακριβώ για απουσία πολιτικής μεροληψίας στην υπόθεση αυτή και σε αυτό είναι κατανοητό και αναγνωρίζεται. Πρέπει να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που αφαιρεί την πολιτική από τι εισαγγελικέ υπηρεσίε. Βέβαια, κανεί δεν είναι ανεξάρτητο. Έχουμε ανεξάρτητε συνεισφορέ, παρεμβάσει εδώ στην αίθουσα, από ανθρώπου που θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητοι, γιατί είναι ακαδημαϊκοί παραδείγματο χάρη. Όμω, οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί που ξέρω εγώ, που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα, μόνο ανεξάρτητοι δεν είναι. Έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για κάτι και είναι τόσο ισχυρή όσο μια άποψη πολιτικού. Έτσι λοιπόν, ε, τώρα από την άλλη, αν μπορούμε να πετύχουμε μια λιγότερο πολιτική εισαγγελία σε όλες τις χώρες, νομίζω ότι θα μπορούσαμε ε, να αντιμετωπίσουμε όλες τις κατηγορίες των εγκληματιών χωρίς φόβο και σε αυτό θα έπρεπε να στοχεύουμε παρά στη συνέχιση αυτής της δύσκολης κατάστασης όπου πρέπει κάποια στιγμή να ληφθούν αποφάσεις για λόγους μη νομικούς και μη καλούς και δεν είναι καλή λόγοι αυτή από άποψη άσκησης δίωξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κερκόπε. Θα ήθελα να σας καθησυχάσω για κάποιες πτυχές. Όσον αφορά λοιπόν την δίκη του Μπερλουσκόνη, ε, κοιτάξτε δεν την έκανε ο κ. Νιούτον Ντάν, την έκανε στη χώρα μου οι δικαστές ε, με πολιτική πίεση. Ε, βέβαια για κάποιες περιπτώσεις καταδικάστηκε, για άλλες ακόμα κατηγορείται. Μπορώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι οι ακροάσεις ε, που οργανώνουμε εδώ, ε, στις ακροάσεις αυτές ε, έρχονται πάντα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και όσον αφορά την ανάκριση και όσον αφορά την δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα πρόβλημα που θα σήμερα να εξετάσουμε. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα που αφορά το ρόλο των τραπεζών ε, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή αυτή στο όλο πακέτο δίμευση. Ο κύριος Ταμπάρευς και μετά η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο συνολικό πανέρμα. Βέβαια, η φορολογική παράδοση είναι πρόβλημα και θα πρέπει να καταργηθούν. Αλλά επίσης πιστεύω πως ε, ε, υπάρχει κάποια διαφορά στον πολιτισμό ε, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ε, σε άλλου και άλλων περιοχών ε, πάνω σε οποίο βασίζεται αυτή η σκιώδης οικονομία και εκεί όχι μόνο χρησιμοποιούνται πόροι που προέρχονται από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες έχουμε κάποιες τράπεζες πάρα πολύ γνωστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δέχονται ε, χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά υπάρχει και διαφορά πολιτισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δημιουργεί τέτοια φαινόμενα, δηλαδή κάτι τέτοιο, τέτοιες αποκλήσεις ουσιαστικά οδηγούν ε, και μάλιστα με την ε, κρίση που είχαμε στις Ηνωμένε Πολιτείε με τα κίνητα μεταφέρθηκαν ε, πάρα πολλά κονδύλια, πάρα πολλά χρήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρωπαϊκό σύστημα. Και σήμερα βέβαια το σύστημα στην Ευρώπη βιώνει όλα αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς η Παγκοσμία Τράπεζα μπορεί να μας βοηθήσει έτσι ώστε να αποτελέσει ένα διάβλο επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών πολιτισμών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, έτσι ώστε να έχουμε ροή των πληροφοριών, επαλήθευση των πληροφοριών και να μπορούμε να επιτρέψουμε όχι μόνο ε, την ε, διήμευση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και μέσω της ανάλυσης διάφορων μοντέλων να προσδιοριστούν πρακτικές ε, που θα είναι πρακτικές καρουσέλ για να διαφεύγει κάποιος την καταβολή φόρων. Αυτή είναι μια πρώτη λοιπόν ερώτηση, πώς μπορεί να βοηθήσει η Παγκοσμία Τράπεζα. Και πιστεύω ότι από τη στιγμή που αυτά τα μεγάλα μπλοκ που προφανώς στο εσωτερικό τους ε, περιλαμβάνουν και σχεδόν φορολογικούς παραδείσους με το μοντέλο που έχουμε στις ΗΠΑ... Πολιτείες όπως το Λουξεμβούργο στην Ευρώπη. Αν ε, όλα αυτά δεν τα επιλύσουμε, βλέπουμε ότι έχουμε και τεράστιες τρύπες σε άλλες χώρες όπως Κίνα, ε, Βραζιλία και τα λοιπά. Χώρες οι οποίες ε, παρόλα αυτά, παρά τα προβλήματα που έχουν στο εσωτερικό τους, ε, ασκούν ε, κριτική, αλλά οι ίδιες δεν καταπολεμούν τις δικές τους γκρίζες ζώνες. Αυτό τώρα είναι ένα σχόλιο που απευθύνεται σε εμά. Δηλαδή, εμεί πρέπει να επιλύσουμε τα δικά μα προβλήματα στι δικέ μα πατρίδε, στο σπίτι μα, για να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον. Και θέλω να ρωτήσω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να ενισχύσουν τη δική τους συνεργασία. Μιλήσουμε εδώ κάπως για τη TFTP. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταπολεμήσει και το οικονομικό έγκλημα και θέλω να ρωτήσω εδώ Ποιο ο συνομιλητή μας συνομιλητής στις Ηνωμένες είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι αυτό που διαχειρίζεται την εφαρμογή της TFTP. Νομίζω ότι ίσω το Κοινοβούλιο εδώ θα έπρεπε να κάνει κάποια δουλειά έτσι ώστε η TFTP να χρησιμεύσει και για την καταπολέμηση του, του οικονομικού εγκλήματο ο κύριος Κίρκοφ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για το FTP και ε, είχαμε, μας είχαν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες, θα πρέπει να μας τις δώσουν και κάποια στιγμή. Ευχαριστώ κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν κατάλαβα που μου κάνατε νόημα. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, με βάση αυτά που είπαν οι συναδελφοί μου, Θέλω να πω το εξή. Όλοι έχουν τα μαρτήματά τους σε όλες οι χώρες. Και η Ιταλία κατά το παρελθόν δημιούργησε προβλήματα. Αλλά και στη δική μου τη χώρα υπήρξαν ε, σκάνδαλα και παρεμπόσεις δικαιοσύνη σε κυρίως σε οικονομικά εγκλήματα, όχι σε ποινικά. Ευτυχώς που εμείς ε, έχουμε τουλάχιστον έναν e e, ευφυή τύπο με σωστές έρευνες που τα προβάλλει όλα αυτά στην κοινή γνώμη. Ε, την ε, ομιλία σας τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί ε, προσθέσατε την πολιτική διάσταση του θέματος που δεν το είχαμε εξετάσει προηγουμένως. Είπατε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι ένας βασικός λόγος γιατί όλα αυτά δεν λειτουργούν και γι' αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να διερωτηθεί που οφείλεται αυτό ε, δέστε ας πούμε Γκαντάφη, Μπερλουσκόνη αλλά και ο Μάρκος ε, στις ε, Φιλιππίνες αυτοί εξαφανίστηκαν και βρήκανε ε, υποστηρικτές ε, που ήθελαν να παρεμποδίσουν την κατάσχεση των ε, περιουσιακών του στοιχείων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αναδυόμενες δημοκρατίες είναι πολύ επιφυλακτικέ και λένε «Μα πού υπάρχει πλέον αυτή η αμεροληψία και η ουδετερότητα». Ε, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ερώτημα. Αυτή η ουδέτερη, αμερόληπτη βάση, πού είναι αυτή. Παλαιότερα υπήρχε η άποψη ότι ο ΠΟΕ και όλα τα άλλα ε, πρόσκυνται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, με εσάς τι γίνεται ακριβώς. Εσείς ε, λειτουργείτε περισσότερο με κανόνες των Ηνωμένων Αθνών ή πώς ακριβώς. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί αυτό μπορεί να είναι και ο λόγος ε, μεγαλύτερης εμπιστοσύνης. Να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι οι κανόνες ε, είναι τα Ηνωμένα Έθνη ε, που θα πρέπει να επικρατούν. Ευχαριστώ πολύ Μπάρμπαρα. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Βαντερντός, αλλά πριν σας δώσω τη λόγο, θέλω να σας πω το εξής, να σας ρωτήσω εξής. Γνωρίζετε ότι στη δική μου τη χώρα σήμερα το πρωί, φρέσκια αυτή τη είδηση, υπήρξαν τράπεζες που κατέσχισαν 4 δις ευρώ από δάνεια ε, που είχαν δοθεί σε μαφιόζους το έκαναν αυτό χωρίς καμία δικαιολογία. Η ε, Barclays ε, κατέσχισε τα χρήματα από παιδιά των μαφιόζων και όταν τους ρώτησαν μα πώς είχε γίνει αυτό να τους δώσετε αυτά τα δάνεια ε, και μιλάμε τώρα για δάνεια που είχαν δοθεί σε παιδιά 20 ετών. Η τραπεζίτες ε, απήντησαν ότι επειδή ήταν παιδιά καλών οικογενειών ε, τους είχαν δώσει αυτά τα δάνεια και γι' αυτό λοιπόν διαρωτώμε πώς είναι δυνατόν όλα να πηγαίνουν στραβά. Στην Ιταλία μιλήσαμε με τέτοιους ανθρώπους που καταγγέλουν το οργανωμένο έγκλημα και αυτοί ζητάνε 15-20 ευρώ δάνειο για να προχωρήσουν, δεν τους δίνουν. Όταν όμως ε, στην περίπτωση όπου ένας 20χρονος ως μαφιόζου ε, ζητά ε, δάνειο 800.000 ε, ευρώ χωρίς καμία έρευνα παίρνει το δάνειο αυτό και απλά και μόνο επειδή θεωρείται ευπρεπές και αξιόπιστο άτομο. Ίσως μπορείτε να απαντήσετε και σε αυτό. Thank you Σας κατευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Πρέπει όμως να φύγω σε ένα τέταρτο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος. Μίλησαν πολύ για φορολογικούς αραδίσους και την χρήση και κατάχρηση τους. Εγώ δεν είμαι ειδικό σε αυτά, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αλλά εδώ στους Puppet Masters στείλτε μου τα στοιχεία σας να σας το αποστείλω, είναι ότι ψάχνουμε ποιο νομικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή αυτοκινήτων ας πούμε που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλες περιπτώσεις και γνωστές διαφθοράς. Νομίζω ότι όχι, μάλλον κάναμε και μια άλλη έρευνα με περίπου 100 εταιρείες που σκεφτόμασταν, που θεωρούσαμε ότι είχαν αποκρύψει χρήματα και θελήσαμε να βρούμε όχι τι θα μας πούν ως πληροφόρηση, αλλά αν μπορούμε να ταυτίσουμε καμία πληροφορία έστω και κρυμμένη. Και πάλι εδώ οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ε, τα κατάφεραν καλά και άρα αυτό που είπε ο κύριος Ταβάρες σημαίνει ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ισότιμη πληροφόρηση, αλλά πρέπει οι πληροφορίες να υπάρχουν καταρχάς. Ότι δεν έχουμε στοιχεία όχι μόνο από τράπεζες αλλά και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καταπιστεύματα σημαίνει ότι υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα γιατί δεν είναι υποχρεωμένα να χορηγούν αυτές τις πληροφορίες ενώ σε άλλες χώρες στην ΣΥΠΑ είναι υποχρεωμένα. Υπάρχει λοιπόν εδώ μεγάλη έλλειψη ισορροπίας αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας για τη γνωστοποίηση των στοιχείων ιδιοκτησίας ή οφέλους. beneficial ownership δηλαδή. British banks with, uh, Και είχε προταθεί κάποτε να εφαρμοστεί ένα, μια σειρά κανόνων για τέτοια πληροφόρηση και χορήγηση πληροφοριών και όταν κανείς είναι συνηθισμένος στη γραφειοκρατική γλώσσα των νομοθετών βλέπει ότι καμιά φορά παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξουν νομοσχέδια που είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Αυτό δεν το λέω για να ψέξω το ή τα β. Ίσα ίσα η έκθεση που ανέφερα ήταν από την Αγγλία και με δημιούργησε, μας προξένησε μεγάλη χαρά. Ποια είστε εσείς κάτω, η κυρία Μάκιντάιρ, α, ναι, ναι. Λοιπόν, για αυτούς που είναι πολύ ισχυροί για να διωχθούν. Αυτό δεν σημαίνει που είπα ότι είναι ευχής έργων αυτό, δυστυχώς είναι γεγονός. Σε πολλές χώρες του κόσμου η δίωξη του πρώην Προέδρου θα δημιουργούσε τέτοια πολιτική διαταραχή ώστε οι κυβερνήσεις συνήθως επιλέγουν να μην το κάνουν. Και γι' αυτό λένε είναι πολύ ισχυρό για να διωχθεί. Γιατί θα δημιουργηθεί τρομερή αναταραχή. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του γεγονότος, αλλά είναι γεγονός. Τουλάχιστον όμως θα έπρεπε οι χώρες να προσπαθήσουν να βρουν τα περιουσιακά του στοιχεία και να τα κατασχέσουν. Αυτό είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν οι χώρες. Την ανάκτηση. Και τώρα για τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία τα πράγματα δεν πάνε καλά διότι 20 με 40 δισεκατομμύρια το χρόνο χάνονται από διαφθορά. Υπάρχει ε, το Asset Recovery Watch όπου προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε για τέτοιες περιπτώσεις και καταλήγουμε σε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια που χάνονται. 5 δισεκατομμύρια πριν από 20 χρόνια. Τώρα είναι όπως σας είπα σχεδόν 40. Τώρα κατά πόσον η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να παρέμβει στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ δεν μπορούμε πράγματι να παρέμβουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όπως λέει και το βιβλίο Puppet Masters είναι να δημιουργήσουμε κάποια ισοτιμία ως προς την συλλογή πληροφοριών. Και για το θέμα των υπερακτίων, όπως λένε στην Κύπρο εταιριών, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν κατάφεραν να βρουν καμία πληροφόρηση. Συνήθως η φορολογική παράδειση αρνούνται, αλλά τουλάχιστον του ζητήθηκε και μπορεί να τρόμαξαν από αυτό. Δεν ξέρω. Αυτή η επιχείρησή μας που την ονομάσαμε Mystery Shopping ε, δεν μας έδωσε στοιχεία. Πρόσφατα ο Jason Sharman, ένας από τους συγγραφείς του Puppet Masters, δημοσίευσε ένα άλλο άρθρο με 2.800 χρηματοπιστωτικές εταιρείες και πάλι το ίδιο διαπίστωσε ότι γενικά δεν απαντούν. όταν ιδίω λειτουργούν σε φορολογικούς παραδείσους ή απαντούν πολύ λιγότερο από ότι οι οργανισμοί σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχει λοιπόν λύση του υπερακτίου προβλήματος αν δεν δούμε και τους παραδείσους. Τώρα για το ερώτημα της κυρίας Βάιλερ, σε ποια βάση γίνεται Question, uh, that we struggle. γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Υπάρχει και άγνοια Συχνά όμως υπάρχει και καχυποψία εκ μέρους των καινούριων κυβερνήσεων. Θεωρούν δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως απριόρι ύποπτα και συνομωτικά. Αφού λοιπόν αυτές οι τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ένοχα γιατί να, μας θέλουν, να θέλουν να μας βοηθήσουν. Και από την άλλη πλευρά αυτά τα ιδρύματα δεν είναι και αυτά σίγουρα μήπως οι αιτήσει δεν γίνονται παρά μόνο και μόνο για πολιτικάντικους λόγους. Μήπως ξαφνικά δηλαδή όλα βγούνε στην πρώτη σελίδα μιας διεθνούς εφημερίδας για να βλάψουν το πιστοτικό ίδρυμα. Υπάρχουν αυτές οι καχυποψίες, ανθρώπινες είναι. Και η μόνη λύση είναι να συνδυαστούν, να συνομιλήσουν τα δύο μέρη και να γράψουν από κοινού την αίτηση, να ε, μοιραστούν τις πληροφορίες και τέτοιου είδους συναντήσεις είναι πάρα πολύ πολύτιμες. Επίσης αν κατάλαβα καλά ρωτήσατε σε ποια βάση δρούμε. Ναι, εδρεύουμε στην Ουάσιγκτον αλλά δεν είμαστε Αμερικανοί και όπως θα δείτε και στο βιβλίο επικρίνουμε πάρα πολύ τις ΗΠΑ για την έλλειψη διάδοσης και χορήγησης πληροφοριών. Δεν λέω ότι δεν κάνουν τίποτα. Ιδιαίτερα αυτοί ζήτησαν περισσότερους κανόνες για πληροφόρηση ιδίως για τα στοιχεία της ιδιοκτησίας και κάποιοι γερουσιαστές ιδίως Δεν λέμε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν έχει αναγνωριστεί στη ΣΥΠΑ, αντίθετα. Το έχουν αναγνωρίσει πάρα πολύ καλά και προσπαθούν να το λύσουν, αλλά για να σας απαντήσω δεν, είμαστε, δεν συνεργαζόμαστε με την Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν είμαστε δηλαδή τμήμα της. Μήπως υπάρχει τίποτε που δεν απάντησα. Νομίζω όχι. Α, ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει μια τραπεζική ένωση. Κάτι που χρειάζεται νομίζω και εδώ χρειάζεται παγκόσμια συνένεση. Καλό είναι να το κάνει η Ευρώπη αλλά άμα δεν το κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος είναι πολύ εύκολο να βάλει κανείς τα λεφτά του αλλού. Πρέπει να είναι λοιπόν και σε αυτό παγκόσμια η στρατηγική. Η ταύτιση αυτού που ωφελείται από την ιδιοκτησία μιας εταιρείας είναι ένας κανόνας που θα έπρεπε επίσης παγκόσμια να εφαρμοστεί για να φανεί αν αν δικαιολογείται η υποψία για χαμηλό δεδηλωμένο εισόδημα και τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό απ' την άλλη. Και εδώ φοβάμαι ότι πρέπει να φύγω. Όμως σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε κύριε Βαντερντός για τις απαντήσεις σας. Όπως είπα και πριν, αν είναι δυνατόν, ε, σας καλώ να αφήσετε την παρουσίασή σας ε, και αν σας έρθει κάποια ιδέα κατά νου ή κάποια περαιτέρω απάντηση, να μας τα γνωστοποιήσετε. Λοιπόν, πριν ε, να φύγουμε, να καταλήψουμε την αίθουσα, θα ήθελα να σας ενημερώσω σε σχέση με την συζήτηση που έγινε με τον Γενικό Διευθυντή κ. Μασερβίση υπήρξε μια σειρά ερωτημάτων. Ίσως ε, τη συζήτηση αυτή θα την ε, ξαναδούμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Αλλά δεδομένη της στρατηγική σημασία των όσων συζητήσουμε και όπως είπε και ο κύριος ε, Μενσερβίς, όσων διακυβεύονται με την οδηγία για τη δίμευση, εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτείτε επί οποιασδήποτε χρήσιμης κοινή δράση που θα μπορούσε να αναλυθεί από αυτή την Επιτροπή γιατί η Κρίμ, ε, η οποία θα έπρεπε να είναι η κόρη της Λίμπε, στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι είναι πολύ πιο αποφασισμένη για αυτά τα θέματα και καθώς αυτό το θέμα είναι κεντρικής σημασίας, εγώ θα σας καλούσα να μην ε, ξεχάσουμε αυτή την τυχή. Παρακαλώ, Βερονίκ. Ίσως να το προσθέσουμε αυτό στην ημερήσια διέταξη για τη συνεδρία των συντονιστών απόψε και να προβλέψουμε για κάποιο χρόνο παραπάνω. Γιατί μάλλον δεν θα προλαβαίνουμε. Πρόεδρος, ναι, βεβαίως, ε, γιατί, όπως είπα, πρέπει να συζητηθεί αυτό το θέμα με τη δεούσα προσοχή, αλλά και αποφασιστικότητα. Παρακαλώ, κύριε Γιαννάκου. Ε, θα σας πρότεινα να οργανώσουμε μια διάσκεψη εδώ στις Βρυξέλλες και να καλέσουμε τους υπουργούς δικαιοσύνης των κρατών μελών. Δηλαδή, να έχουμε άμεση επικοινωνία, άμεση επαφή με τους υπουργούς δικαιοσύνης. Θα ήταν μια καλή ιδέα. Συμφωνώ μαζί σας. Και για μένα λοιπόν Κοιτάξτε, είπα ότι συμφωνώ μαζί σας, θαυμάσει αυτή η ιδέα. Θα ενημερώσουμε ε, τους συντονιστές ε, για αυτό το θέμα, για αυτή την πρόταση. Και ο Διευθυντής Μανσερβίση μας είπε ότι ε, είναι προνομία του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Αλλά και εμείς προχώμαστε από κράτα μέλη. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν πρωτοσυστήθηκε αυτή η Επιτροπή, πολλοί συνάδελφοι ε, με ρώτησαν ε, μήπως ε, εγώ ή εσείς θα θέλατε να οργανώσουμε συνέδρια στα κράτη μας και αυτό για να ευαισθητοποιήσουμε τις κυβερνήσεις μας. Να ευαισθητοποιήσουμε τους ομόλογους μας, τους συναντέλφους πολιτικούς στα κράτη-μέλη. Εγώ έχω απόλυτη ευθύνη για όλη αυτή την υπόθεση. Πρέπει όμως να σας πω ότι τελικά δεν έγινε τίποτα. Εκεί σταμάτησε. Δηλαδή τον προηγούμενο μήνα πήγα στη Γερμανία, στην Κολονία και συμμετείχα μεταξύ άλλων σε μια πολυπληθέστατη συνάντηση ε, και δεν ήταν ε, μόνο δικαστές και ανακριτές, ε, ήταν μια ανοιχτή συζήτηση στην κοινωνία των πολιτών και όλοι αυτοί ήθελαν να καταλάβουν, να κάνουν ερωτήσεις, επιθυμούσαν να γνωρίζουν. Ε, υπάρχει λοιπόν μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρου των ε, αρμόδιων αρχών και των πολιτικών των κρατών μελών. Και όχι διότι δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου στα κράτη-μέλη. Υπάρχει δηλαδή αφενός ε, η πολιτική βούληση, η οποία όμως ε, λέει ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά οι πολιτικοί δυστυχώς δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν εναπόκειται σε εμά να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί να καταστήσουμε για άλλη μια φορά σαφές στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο δεν θα είναι πια παθητικό <clears throat> αλλά είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στο θέμα αυτό. Θα ξανασυζητήσουμε λοιπόν το θέμα στις συνεδρίες των συντονιστών και σας υπενθυμίζω ότι θα ξεκινήσουμε στις 3 ε, ε, και στις 5.30 ε, θα έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Καλή σας όρεξη.